Ας ξεκινήσουμε. Βέβαια δεν έχουμε εδώ τον εισηγητή για να ξεκινήσουμε. Can somebody ask where Mrs. Η κυρία Τρύπελ, ξέρετε που βρίσκεται. Good morning. I am, starting... Καλημέρα. Θα ξεκινήσω με κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα καταρχήν να σας ζητήσω να διαβάσετε προσεκτικά τις αποφάσεις των συντονιστών. Θα τα λάβατε σίγουρα ηλεκτρονικά. Ε, αν έχετε κάτι να πείτε, σας παρακαλώ πολύ, στο τέλος της συνεδρίασης να το πείτε, γιατί πρέπει να εγκριθεί να εγκριθούν οι αποφάσεις των συντονιστών και πρέπει να το κάνουμε στο τέλος συνεδρίας. Κυρία Τρούπελ, βλέπω να έρχεται, καθίστε, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως με τις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε. Προϋπολογισμός 2010. Έχουμε τροπολογίες. Η Χέλγα θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες για τις τροπολογίες. Καλημέρα σε όλους. Όσον αφορά τις γενικές ε, παρατηρήσεις, ξέρετε ότι τους πόρους οι οποίοι είναι στη διάθεσή μας, όπως ακούσαμε χθε και από την Οντίλ Κοντά που μας ε, έκανε την παρουσίαση, δεν αρκούν. Οι πόροι δεν αρκούν. Και το 2010 καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε πλήρως να παίξουμε το ρόλο μας. Όταν όμως γίνει η συζήτηση για την αναθεώρηση, η γενική συζήτηση για τον προπολογισμό, σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να εκφράσουμε τις προτεραιότητές μας και να πούμε και πού θέλουμε να δοθούν οι προτεραιότητες. Τα κονδύλια για τα μέσα, τα οπτικοακουστικά, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση δεν αρκούν. Στη γενική συζήτηση λοιπόν η οποία πρέπει να γίνει θα ε, εκφράσουμε αυτήν την θέση μας, αυτήν την απέτησή μας και ελπίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ε, θέμα αυτό θα μπορέσουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στις δικές τους εθνικές κυβερνήσεις. Τώρα, προϋπολογισμός 2010. Προσπαθήσαμε παρόλο τον περιορισμό των κονδυλίων να δώσουμε έμφαση σε κάποιους τομείς, παραδείγματος χάρη πολιτική στον τομέα της επικοινωνίας, networking. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις, συνεργαζόμενοι στενότερα με τους δημοσιογράφους, με τα κανάλια, με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, όχι μόνο στις προεκλογικές ε, περιόδους, αλλά πάντα και συνεχώς. Επίσης, ε, Προσπαθήσαμε να δοθούν περισσότεροι πόλεις στο Εράσμους και σε άλλα προγράμματα τα οποία γνωρίζουν πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε προγράμματα και θέματα και μηνύματα τα οποία γνωρίζουν οι νέοι, γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα οποία τους φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά. Δηλαδή προγράμματα για την εκμάθηση των γλωσσών, για την ανταλλαγή σπουδαστών, κάτι που αυξάνει την ευρωπαϊκή συνείδηση των νέων. Και άλλα πολύ σημαντικά σημεία για την δική μας πολιτιστική πολιτική, πιλωτικά προγράμματα, που όπως ξέρετε ήδη από την πρώτη ανάγνηση προσπαθήσαμε να προωθήσουμε το θέμα του cross-border των δημοσιογράφων και στην πρώτη ανάγνωση και την πρώτη συζήτηση εξάλλου που ε, είχαμε για το θέμα αυτό υποβλήθηκαν διάφορες τροπολογίες. Τις περισσότερες τις ε, στηρίζω. Πρόκειται για αποσαφηνήσεις, για καλύτερη διατύπωση. Ένα σημείο δεν μπορώ να δεχτώ. Οι άλλες τροπολογίες με τις οποίες δεν συμφωνούσα αποσύρθηκαν. Πιστεύω ότι η σημερινή ψηφοφορία δεν μπορεί παρά να είναι αρμονική γιατί υπήρξε προηγούμενη συμφωνία για τις περισσότερες τροπολογίες. Πρόεδρος, νομίζω ότι η συζήτηση έγινε, δεν θα την επαναλάβουμε. Η κυρία Παλιαντέλη Δεν είναι εδώ, αλλά ξέρω ότι υπήρχε κάποια αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, ψηφίζουμε. Έχετε όλοι τον κατάλογο. Απαρτία υπάρχει. 9 από το ΕΛΚ, 5 από τους σοσιαλιστές, 2 από τους πράσινους, 2 από τους ε, τιγκούε και ένας από τους φιλελεύθερους. Α, και ένας μη εγγεγραμμένος. Έχετε τον κατάλογο. Ψηφίζουμε την παράγραφο 1, τροπολογία 1 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 2. Κώστα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Τροπολογία 3. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Τροπολογία τέσσερα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4α. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Παράγραφος 5 και τροπολογία 8. Υπέρ. Μετράμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 6α. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6α. Αποσύρθηκε. 6γ. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6α, τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6α πάλι, πρόκειται για την 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Χρειαζόμαστε και τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Τρούπελ. κατά αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τρούπελ. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο σημείο της ε, σημερινής ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για το σημείο 9 και πρόκειται για το Ευρωπαϊάννα. Τα επόμενα βήματα. Στις 2 Σεπτεμβρίου η Έλγα Τρούπελ ορίστηκε σαν εισηγήτρια για την έκθεση αυτή και όλοι γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό είναι ένα online ε, βιβλιοπωλείο, είναι ένα είδος αρχείου. Το 2008, το Νοέμβριο, άνοιξε σαν τμήμα της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη η πολιτιστική κληρονομιά και η λογοτεχνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο έχει σημασία και για το μέλλον και βεβαίως, όπως ξέρετε, πολύ σημαντικά θέματα μας αφορούν. Πρώτον, το περιεχόμενο. Τι μπορεί κανείς να δει σε αυτό το Ευρωπαϊκό. Δεύτερον, η οργάνωση ποιος πληρώνει, ποιος έχει την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και τα λοιπά. Η κυρία Τρίπελ σίγουρα θα έχει επεξεργαστεί το θέμα αυτό και θα έχει και κάποιες πρώτες προτάσεις σε γενικές γραμμές το θέμα αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητήσαμε χτες όσον αφορά την πρόσβαση στο Google και την ψηφιακή παρουσίαση των βιβλίων. Επίσης το θέμα του copyright, των πνευματικών δικαιωμάτων και επουδενή λόγο δεν πρέπει να δώσουμε ένα λάθος μήνυμα ε, για το θέμα αυτό. Η κυρία Τρίπελ στις 30 Νοεμβρίου θα είναι έτοιμη για να υποβάλει την εκθέση της και τώρα απλώς θα ακούσουμε κάποιες πρώτες ιδέες και σας παρακαλώ αντιδράστε έτσι ώστε να ακουστούν οι απόψεις σας, οι αντιδράσεις σας και να μπορέσει η κυρία Τρίπελ να τη συμπεριλάβει στην έκθεσή της. Χέλγα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Την τελευταία νομοθετική περίοδο ξεκίνησε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ήμασταν τότε στην φάση προετοιμασίας της, ε, του Ευρωπαϊάνα. Λήφθη κατά κάποιο τρόπο η πρώτη απόφαση και υπήρξε συμφωνία για τη δημιουργία ενός μεγάλου ε, φιλόδοξου σχεδίου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη. Συζητήσαμε αμέσως βεβαίως και θέματα προεπολογισμού και πρέπει να σας πω ότι δεν συνεργαζόμαστε μόνο με μεγάλους ε, φορείς του διαδικτύου όπως το Google, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ψηφιακή ενσωμάτωση αυτών των έργων δεν είναι πάντα κάτι που γίνεται από το Google. Υπάρχει το πρόγραμμα του Google, το e-book settlement, και το θέμα είναι τα δικαιώματα των συγγραφέων αυτών των βιβλίων, γιατί πολλές φορές ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δικαιώματα των ε, συγγραφέων αυτών που είναι ακόμα στη ζωή, που είναι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν ε, διέθεσαν στο διαδίκτυο μόνο βιβλία τα οποία ήταν εκτός copyright. Γι' αυτό και συζητήσαμε το θέμα αυτό στη φάση αυτή προετοιμασία. Το αμερικανικό copyright είναι κατά κάποιο τρόπο πιο ευάλωτο. Στην Ευρώπη υπάρχει η λεγόμενη fair use, η χρήση δηλαδή, η οποία κατά κάποιο τρόπο μας επιτρέπει να παρεκκλίνουμε από το copyright. Αντίθετα, στην Αμερική είναι πολύ πιο ε, δύσκολη η κατάσταση, γιατί το, οι συγγραφείς, όπως ξέρετε, έχουν μια προστασία η οποία είναι πολύ πιο δύσκολο να παρακαμφθεί. Είχαμε λοιπόν στην πρώτη φάση προετοιμασία συναντήσεις με εκδότες, με εκδοτικούς οίκους, με συγγραφείς, και με ειδικού για την ψηφιακή διάθεση των έργων στο διαδίκτυο. Η κεντρική ιδέα ήταν πιο εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά προστασία και δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Δηλαδή, σκοπός μας είναι να υπάρχει ελεύθερη ή εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ε, οικονομική επιβάρυνση. Δεν είναι δωρεάν. Στην ε, Σουηδία και στην ε, Γερμανία συζητήσαμε και με αυτούς οι οποίοι ονομάζονται πειρατές. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δούμε πώς τα δικαιώματα παρόλα αυτά θα προστατεύονται, ενώ ο αρχικός σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να υπάρχει διαθέσιμο υλικό στο διαδίκτυο. Τα περιεχόμενα αυτών των βιβλίων, λοιπόν, ε, και αυτή είναι η κεντρική ιδέα, θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Αυτοί όμως οι οποίοι ζουν από αυτήν την εργασία και οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα σε πνευματικά δικαιώματα, αυτό δεν θα πρέπει να καταρρεύσει επειδή τα έργα τους είναι πλέον διαθέσιμα στο ίντερνετ. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, ξέρετε ότι υπάρχει όλη αυτή η κοινότητα του ίντερνετ και η πειρατές του κυβερνοχώρου, όπως τις ονομάζουμε, οι οποίοι βεβαίως έχουν ε, την εντύπωση ότι πρόκειται για εμπόδιο στην ελεύθερη διάδοση της γνώσης και της δημιουργικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο, ο οποίος να διαθέτει μεν τα προϊόντα αυτά, αλλά να προστατεύει τα δικαιώματα των ε, συγγραφέων δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη μία και μοναδική διάθεση. Κάθε φορά που υπάρχουν αντίγραφα δεν μπορεί να ζητούνται πνευματικά δικαιώματα. Εξετάσαμε λοιπόν όλες αυτές τις περιπτώσεις και με την κυρία Κοντά προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες ε, ε, δυνατότητες να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και να διαθέσουμε το υλικό αυτό με έναν τρόπο που να μην εμποδίζει τη διάθεσή του. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και πρέπει να σας πω ότι χρειαζόμαστε ακόμα πολλές ιδέες τεχνικές αλλά και πολιτικές για την ε, πρόθεσή του. Το 2008 ξεκίνησε το Ευρωπαίνα με έναν πρώτο κατάλογο των έργων. Η Γαλλία, αν θέλετε, είναι πρώτη σε αυτόν τον κατάλογο γιατί έχει ήδη περάσει σε ψηφιακή γλώσσα τα περισσότερα έργα στην Ευρώπη, 10% περίπου, και κατόπιν ακολουθούν άλλες χώρες. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο εύκολα προσβάσιμη. Τι έκανε μέχρι τώρα το Ευρωπαίανα και το οποίο θεωρώ και πάρα πολύ σωστό, βιβλία εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε έργο, είτε πρόκειται για βιβλίο, είτε πρόκειται για κάτι άλλο, το οποίο είναι ακόμα copyright και για να μην υπάρχει μεγάλο κενό στα έργα του 20ου αιώνα, πλησιάσαμε όλες τις αρχές, τις αρμόδιες αρχές ή τους συγγραφείς, αν είναι ακόμα εν ζωή, οι οποίοι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα και κάναμε τις αιτήσει για να μπορέσουν να διατεθούν τα έργα αυτά στο διαδίκτυο. Ξέρετε ότι το Αμερικανικό Δικαστήριο, το οποίο έχει επιληφθεί αυτής της υπόθεσης, των copyright, στις 7 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει την εξέταση του θέματος. Στις 6 Νοεμβρίου οργανώνεται μια μεγάλη ακρόαση στην Αμερική για το θέμα αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων και τη διάθεση των έργων με ψυχιακή μορφή στο διαδίκτυο. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όλους μας και για το Ευρωπαϊκό. Καταλαβαίνετε ότι μιλώντας για το Ευρωπαίανα, συζητήσαμε για θέματα πολύ πιο γενικά. Παραδείγματος χάρη αν το θέμα αυτό θα ρυθμίζεται από κάποιες κεντρικές αρχές, κρατικές ή ευρωπαϊκές, ή αν θα είναι ένα άλλου είδους ε, μοντέλο. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει κονδύλια. Πριν από λίγες εβδομάδες οργανώθηκε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα, μια ακρόαση, η κυρία Ρέντινγκ ήταν παρούσα, ακολούθησε μια συνέντευξη τύπου όσον αφορά τις τεχνικές δυνατότητες αλλά και τα κονδύλια που χρειάζονται. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν μία δημόσια αρχή, ευρωπαϊκή αρχή, θα μπορέσει να αναλάβει και να πλαισιώσει όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε στο Google όλη την ε, ανάπτυξη αυτού του σχεδίου. Η κυρία Ρέντιν, κατά την άποψή μου, βιάστηκε. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο ε, έτοιμη να εγκαταλείψω την προσωπική μας θέση, η οποία σαφώς και είναι η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης να ρυθμιστεί από εμάς γιατί δεν μπορούμε τα πνευματικά αγαθά αυτά, τα οποία αποτελούν τον πολιτισμό της Ευρώπης, να τα ε, εγκαταλείψουμε και να τα αφήσουμε ελεύθερα, χωρίς καμία, ε, αν θέλετε, προϋπόθεση και όρο. Ε, είμαι σίγουρη ότι και στην Αμερική το θέμα αυτό έχει πάρει τέτοια ε, δημοσιότητα και τέτοια σημασία που δεν πιστεύω ότι θα το εγκαταλείψουν ε, χωρίς όρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν τις απόψεις για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μάτιν ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Την εισηγήτρια. Εξαιρετικά σημαντικό το θέμα, ε, υψηλή σημασία, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η μέχρι τώρα δουλειά που έχετε κάνει. Εδώ και πολλά χρόνια Äh, die bequem davon leben können, auch was Sie zum Thema Wissengesellschaft gesagt haben. Πιστεύω που έχει φτάσει, αν θέλετε, η διάδοση του ίντερνετ στους νέους, δεν πρέπει που λόγο να δώσουμε την εντύπωση ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε το περιεχόμενο και τις γνώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα σωστό μήνυμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό θα πρέπει λοιπόν να είναι προσεκτικοί. Και έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Εγώ είμαι νέο μέλος αυτής της Επιτροπής. Υπάρχουν εναλλακτικέ δυνατότητες χρηματοδότησης. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το Google, τι άλλες πηγές χρηματοδότησης ε, ενδεχομένως μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί έχουμε αυ το Google, που είναι ένας μεγάλος αμερικανικός ε, φορέας, ενεργός και παντοδύναμος στο ίντερνετ, αλλά τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν. Άλλη ερώτηση. Μία ευρωπαϊκή εγκυκλοπαίδεια, Ευρωπαίανα θα μπορούσε να δημιουργηθεί και στην Αυστρία αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε πολύ πλούσιες βιβλιοθήκες, εθνικές βιβλιοθήκες και δεν μπορούν τα κράτη από μόνα τους να κάνουν μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Πώς ε, βλέπετε αυτήν την ιδέα, όπως την παρουσίασε η κυρία Ρέντινγκ με το Google, υπάρχει κάτι το εναλλακτικό που θα μπορούσαμε εμείς να προτείνουμε. Και πιστεύω ότι με τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε σήμερα, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να υποβάλουμε ήδη κάποιες πρώτες ιδέες έτσι ώστε να διαδοθούν, να γίνουν γνωστές και να στηριχτούν από το ευρύ κοινό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Του. Euh, euh, Ευχαριστώ, Helga, για τα όσα είπατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα ήθελα να φέρω στη συζήτηση το θέμα των ανθρώπων που έχουν δυσκολίες ε, γραφής. Ε, που έχουν πρόβλημα όρασης, είναι τυφλοί ή αναλφάβετοι ή νέοι οι οποίοι δεν έχουν πάει στο σχολείο αρκετά. Προβλέπετε κάτι για τους ανθρώπους που έχουν δύσκολη πρόσβαση στην γραφή. Για παράδειγμα στη Γαλλία αυτό που φτιάχνουμε είναι CD, CD. CD δηλαδή με ηθοποιούς που διαβάζουν τα κείμενα για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο γραπτό κείμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούρια. Ευχαριστώ. Εγώ συμμερίζομαι τα όσα είπε η κυρία Τρούπελ για την δυνατότητα να βρούμε έναν συνομιλητή στον δημόσιο τομέα. Πέρα λοιπόν από τα όσα προβλέπονται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο μας έχει κάνει ένα απολογισμό, ένα μάλλον υπολογισμό για το πόσους πόρους χρειάζεται για να μπορούμε να δούμε ποιος μπορεί να στηρίξει αυτή τη δαπάνη ή αν υπάρχουν και περισσότεροι από ένας που μπορούν ε, ίσως να στηρίξουν αυτή τη δαπάνη. Επίσης, συμμερίζομαι και την παρατήρηση της ε, προλαλήσασης, γιατί κατά την άποψή μου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα, επειδή είμαστε η Ευρώπη, να μπορέσουμε εδώ να συμμετέχουν και άτομα με ειδικές ανάγκες ή που έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση στην ε, ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τη συνάδελφο για τις τόσο καλές επεξηγήσεις που μας έδωσε για το θέμα αυτό. Ίσως και είναι το πιο σημαντικό θέμα που έχουμε επιτάπητος εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού που συμπεριλαμβάνει τις νέες τεχνολογίες και την στήριξή μας στους δημιουργούς. Όχι μόνο του Ευρωπαίαν αλλά γενικότερα και στο διαδίκτυο. Αναφέρθηκε η σουηδική περίπτωση των ε, πειρατών του κυβερνοχώρου. Νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο πολύ ζωντανό σε όλες τις χώρες και στην Ισπανία. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες όπου οι νέοι κάνουν τέτοιου είδου πειρατεία εντό αγωγικών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι οι νέοι πολλές φορές δεν νιώθουν ότι κάνουν κάτι που δεν πρέπει, Κάποιο ο οποίο κλέβει, α πούμε, ένα μήλο από ένα σούπερ μάρκετ είναι αλλιώ. Το να κατεβάσει κάτι από το διαδίκτυο δεν το βλέπει σαν κάτι κακό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Και η δικιά μα επιτροπή, αλλά και άλλε, οι νομικοί, οι βιομηχανία, έχουν ευθύνη για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Δεν λέω ότι υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή, ώστε να συνδυαστούν οι νέες τεχνολογίες με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά να το Ευρωπαϊκό είναι ένα παράδειγμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις εκτός Google και ίσως και εκτός ε, δημοσίων οργανισμών. Στη Μαδρίτη έχουμε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά τον πολιτισμό, από όποιο επίπεδο και αν το δούμε δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν σημαντικό η Επιτροπή μας να καθίσει και να συζητήσει το θέμα των σπόνσορ, ε, των ε, ανθρώπων ε, που μπορούν να προσφέρουν χρήματα για να στηρίξουν τη δημιουργία, τον αθλητισμό. Να βρούμε δηλαδή με εκείνες που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά να δούμε τι ισχύει για αυτό το θέμα στις διάφορες χώρες και να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Να συγκρίνουμε μάλιστα τι ισχύει στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Αμερική. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο για μας και για τις επιχειρήσεις, τους μεκίνες, να είναι κάτι ξεκάθαρο, τι κανόνες δηλαδή ισχύουν στην περίπτωση που προσφέρουν χρήματα για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Κυρία καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί για μια πρώτη παρουσίαση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Πιο εύκολη πρόσβαση στη λογοτεχνία, στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Υπάρχουν πολλά έργα που με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν ε, πιο γνωστά και πολύ πιο εύκολο να τα γνωρίσει κανείς. Πιστεύω ότι δεν πρέπει που δεν είναι λόγο να υποτιμήσουμε το μέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης αυτό που είπε η συγγήτρια, το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το θέμα όπως το έκανε το Google, δηλαδή αγνοώντας πλήρως το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και της προστασίας των δημιουργών. Ε, διότι όπως ξέρετε δεν μιλάμε μόνο για λογοτεχνία, μιλάμε για καλλιτέχνες ε, των οποίων η δημιουργία προϋποθέτει ε, δαπάνες. Και δεν υπάρχει τέχνη χωρίς έξοδα, χωρίς δαπάνες, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Είναι αδύνατον να μην λάβουμε υπόψη μας αυτό σαν πρωταρχικό δεδομένο, ε, ιδιαίτερα όταν απευθυνόμαστε σε νέους. Πιστεύω ότι για τους νέους χρειάζεται όντως ευαισθητοποίηση. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι η πρόσβαση στον, στο διαδίκτυο δεν μπορεί να γίνεται μόνο δωρεάν και αυτό είναι κάτι που τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες θα πρέπει να το συζητήσουμε σε πολλούς τομείς. Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα το βρούμε μπροστά μας μόνο στη συζήτηση για το ευρωπαίανα Έχει συνέπειες και σε πολλούς άλλους τομείς, ε, όσον αφορά παραδείγματο χάρη την τέχνη γενικότερα, τον κινηματογράφο και γι' αυτό και πιστεύω ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού θα πρέπει να δούμε τις πηγές χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος και αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης, ένα τέτοιο ε, σχέδιο θα πρέπει να στηριχθεί και από τον ιδιωτικό τομέα και από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Είναι τόσο σημαντικό που θα πρέπει να το παρουσιάσουμε ευρέως. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας ε, για αυτό το θέμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και εμπίπτει στην ισορροπία των προτάσεων ανάμεσα στα πνευματικά δικαιώματα και τα καταναλωτικά δικαιώματα. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο για τα δικαιώματα αυτά και για την ε, διάδοση των πληροφοριών και την πρόσβαση στη τέχνη και τη λογοτεχνία. αναγνώριση των καλλιτεχνών και η οικονομική τους ανταμεβή είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και ευκαιρίες όπου οι καλλιτέχνες ήδη θα μπορούν να πούν σε ποιο βαθμό θέλουν να ανταμειχθούν οικονομικά, διότι υπάρχουν κάποιες ε, μέθοδοι όπου οι καλλιτέχνες μπορούν, για παράδειγμα, να δίνουν τα δικά τους προϊόντα δωρεάν, διότι θεωρούν ότι μπορούν οι ίδιοι να ωφεληθούν από τη μεγαλύτερη διάδοση της παραγωγής τους ε, ή της ε, δωρεάν πρόσβασης σε αυτήν. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει αυτό να το δούμε σε αντίθεση με τα εμπορικά δικαιώματα που μπορεί να οδηγήσουν αυτή τη συζήτηση πέρα από τα πραγματικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα των ε, καλλιτεχνών. Θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή και την ισορροπία ανάμεσα στα πραγματικά δικαιώματα και τα καταναλωτικά δικαιώματα. Ich will die Kollegen nur daran erinnern, wir reden jetzt nicht θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να συνειδητοποιήσετε ότι το θέμα του copyright των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ευρύτερο. Θα το συζητήσουμε πολλές φορές ακόμα και στα πλαίσια και άλλων θεμάτων. Ας μην επικεντρωθούμε λοιπόν μόνο σε αυτό το θέμα. Ας συγκεντρωθούμε στο Ευρωπαϊνά, που είναι το σημερινό μας θέμα, και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, του copyright, θα δείτε ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να το ξανασυζητήσουμε. Θα οργανώσουμε μια ακρόαση κοινή με την νομική επιτροπή. Θα είναι, αν θέλετε, το θέμα του 2010, το copyright. Η κυρία Καμαέβαρτ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τρίπελ. Καταρχήν συμφωνώ με τις δύο μεγάλες κατευθύνσεις όπως μας τις προτείνετε όσον αφορά δηλαδή την ελεύθερη πρόσβαση που δεν σημαίνει δωρεάν. Αυτό είναι μια ιδέα που δεν πρέπει να την ε, εγκαταλείψουμε. Ε, το θέμα είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, μέχρι πού θέλουμε να τα προστατεύσουμε. Παρόλα αυτά η ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης ή εύκολης πρόσβασης σε χαμηλό κόστος και της προστασίας των δημιουργών είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς μπορούμε δηλαδή να διαθέσουμε ένα βιβλίο ε, χωρίς αυτό να εμποδίζει, αν θέλετε, την ε, πρόσβαση δεν μπορεί να γίνει δωρεάν σίγουρα, αλλά θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που οι νέοι να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Και την ίδια ώρα επαναλαμβάνω να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης και της προστασίας των ε, καλλιτεχνών, των συγγραφέων, των δημιουργών. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε έναν κεντρικό ευρωπαϊκό φορέα, ο οποίος θα ασχοληθεί και θα πλαισιώσει όλη αυτή την προσπάθεια διάθεσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Γιατί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι κάτι που θέλουμε να προστατεύσουμε και να το διαθέσουμε σε περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες. Όντως χρειάζεται να σκεφτούμε νέους τρόπους συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ακούσαμε την ανακοίνωση της Επιτροπής θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δυνατότητες των κρατών μελών, εκδοτική ήχη και ένας τρόπος χρηματοδότησης ίσως θα μπορούσε να είναι και μέσω της διαφήμισης. Δηλαδή, γιατί να μην το σκεφτούμε και αυτό. Μιλάμε για πολιτιστική χρηνομιά και ενδεχομένως δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαφήμιση, ίσως μέσω της διαφήμισης των κινητών, των απορριπαντικών. Τι να σας πω, πρέπει να προσέξουμε πώς θα το χειριστούμε το θέμα αυτό. Εδώ στην έκθεση διαβάζω ότι όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των ε, έργων τέχνης, θα πρέπει να υπάρχει παρόλα αυτά κάποιο δικαίωμα πρόσβασης. Δηλαδή, ακόμα και για τα έργα των οποίων το copyright έχει πλέον πάψει να ισχύει, εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ε, κόστος για τους χρήστες. Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν ξέρω αν στέλνουμε το σωστό μήνυμα προς τα έξω, αν ακόμα και για παλιά έργα ζητάμε κάποιο δικαίωμα πρόσβασης. για βιβλία παραδείγματο χάρη κλασικά του 1800. Έχω την εντύπωση ότι στην Ευρωπαϊκή θα πρέπει να επιλέξουμε σωστά καταρχήν τα βιβλία τα οποία θέλουμε να διαθέσουμε. Γιατί δεν ξέρω αν οι νέοι σήμερα ενδιαφέρονται τόσο πολύ για βιβλία φυσικής ιστορίας ή επιστημονικά συγγράμματα του 1893, όπως είδα ότι έχουν συμπεριληφθεί στους καταλόγους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ την εισηγήτρια για την παρουσίασή της. Θα ήθελα επίσης να επικεντρωθώ λίγο στις εμπορικές πτυχές Ακούσαμε τις ανησυχίες όσον αφορά το Google. Αν δεν υπάρξει δράση άμεσα, θα καταλήξει σε ένα εμπειρικό εγχείρημα. Και εγώ νομίζω ότι κάτι λείπει εδώ στο ευρωπαϊκό σύστημα με το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν ιστορικές αξίες. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ψηφιακή μορφή σε περιεχόμενο, το οποίο έτσι δεν υπάρχει σε καμία άλλη μορφή. Και δεν μιλάω μόνο για τις πιο πρόσφατες ε, παρουσιάσεις, αλλά και για πιο παλιές, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να φροντίσουμε οι αξίες αυτές, το, η αξία αυτή των εκδόσεων να παραμείνει. Το Google δεν ξέρουμε τι αξία έχει, γιατί η αξία αυτή των ψηφιακών μέσων δεν ε, μας επιτρέπει να πούμε ότι τα βιβλία αυτά θα παραμείνουν. Η πολιτιστική πτυχή δηλαδή είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν θα πρέπει να βασιστούμε μόνο στο Google. Θα ήθελα επίσης να τονίσω και μια άλλη πτυχή. Όπως και να χειριζόμαστε το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και όπως και αν επιτρέπουμε να χρησιμοποιείται αυτή οικουμενικά, νομίζω ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κάπως πιο εμπορικό εκ παραλίλου. Δηλαδή παρά αυτή την δημόσια πτυχή που δίνουμε στα αρχεία μας, λέμε πρόσβαση στα δεδομένα μας, πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί συγχρόνως το Google λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Τα πλεονεκτήματα ε, που δίνουν είναι πολλά. Εμείς είμαστε κάπως πίσω, έχουμε μείνει πίσω. Γι' αυτό και θα ήθελα να προσπαθήσουμε τα εθνικά συστήματα να γίνουν πιο γρήγορα. Ο αρμόδιος επίτροπος θα έπρεπε να φροντίσει για τον έλεγχο αυτών των εθνικών συστημάτων, εννοείται να είναι συμβατά μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην καθυστερούμε πολύ και να μην μένουμε τόσο πολύ από το Google. Να ελέγξουμε δηλαδή την μετατροπή σε ψηφιακά δεδομένα του υλικού που διαθέτουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Και εγώ συμφωνώ με τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσης αυτής. Μια υπόθεση όπως το Ευρωπαϊκά, όπως και άλλες που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, μας κάνουν να αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε αλλιώς. Αναγκαζόμαστε λοιπόν ε, να σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο μέσα στα σύνορά μας, αλλά δεν υπάρχουν σύνορα για το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα μέσο το οποίο βέβαια μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες συγχρόνως. Τρία πράγματα θέλω να θίξω από το θέμα αυτό. Πρώτον, η σημασία που έχει προστασία των δημιουργών, των συγγραφέων. Ο κίνδυνος που υπάρχει για να χαλάσουν όλα αυτά και η προστασία του, της πολιτισμικής διάστασης. Βρισκόμαστε σε μια δεδομένη κατάσταση, μην το ξεχνάμε, και ξέρουμε ότι δεν έχουμε αρκετά μέσα. Αυτό πλήττει τομείς κυρίως όπως είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Ψηφίσαμε τον προπολογισμό, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Ακούσαμε χθε την κυρία Καντά η οποία μας είπε ότι για πολλούς τομείς δεν είχε αρκετά χρήματα στη διάθεσή της για να προχωρήσει. Ακόμα και αν δεν το είπε έτσι ομά, νομίζω ότι αυτό υπονοούσε. Μάλιστα ανησυχώ ακόμα περισσότερο για τέτοιου είδους θέματα, γιατί όταν δεν έχουμε χρήματα για αυτά, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι το θύμα. Είναι τελικά εκείνοι οι οποίοι έχουν περισσότερες δυσκολίες να έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους τα σύγχρονα μέσα. Αυτοί λοιπόν πλήττονται πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ φοβάμαι ότι φτιάχνουμε μια κοινωνία πολλών ταχυτήτων. Ό,τι και αν κάνουμε, πράγματα όπως το Google ε, αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και το περιεχόμενο του Ευρωπαίανα και πώς ευνούμε την πρόσβαση σε τέτοιου είδους μέσα. Είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά κάτι το εξαιρετικό. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες εδώ, κοινωνία πολλών ταχυτήτων. Με το Ευρωπαίανα πρέπει να δούμε τη ρύθμιση. Το Google ό,τι και να κάνουμε εμείς θα προχωρήσει θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Βλέπουμε και στην Κίνα τι γίνεται. Τι δυναμικό υπάρχει εκεί οικονομικά στην Κίνα. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν μέτρα ρύθμισης. Έπειτα συμφωνώ με τη δικιά σας την ανάλυση για τους κινδύνους που υπάρχουν να είναι όλα δωρεάν. Ναι, αλλά αν δεν είναι όλα δωρεάν, τότε πόσο θα κοστίζουν, ποια θα είναι η τιμή είναι πολύ βασικό να καθίσουμε να σκεφτούμε πάνω σε αυτό, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την βιβλιοθήκη. Η τιμή δηλαδή να μην είναι αποτρεπτική, να μην καταλήξουμε σε αυτή την κοινωνία πολλών ταχυτήτων, αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μέσο το οποίο είναι και παιδαγωγικό, έτσι, εκπαιδευτικό. Πολύ ωραίο. Αυτοί που δεν έχουν τα μέσα, τι θα κάνουν, δεν θα απευθυνθούν σε άλλα μέσα τα οποία κινδυνεύουν να έχουν όλα τα αρνητικά που αναφέρθηκαν πριν. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της προστασίας των δεδομένων επίσης και άκουσα κάποιες παρεμβάσεις πάνω σε αυτό για το πώς δηλαδή οι νέοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σήμερα. Εμείς εδώ είμαστε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να φροντίσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους νέους κυρίως, να τους ενημερώσουμε για τους κινδύνους που υπάρχουν από τη χρήση του διαδικτύου μερικές φορές. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι μόνο. Εάν η Επιτροπή μας προσφέρει να πάρουμε κονδύλια από την πολιτική της επικοινωνίας, τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δηλαδή από το προϋπολογισμό της Βάλστρουμ. Καλή ιδέα, δεν σας φαίνεται αυτό. Να το ξανασκεφτούμε. Κυρία Παλαντέλη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ την κυρία Τρίπελ για, τα, για όσα μας είπε σχετικά με την Ευρωπαϊκή και βέβαια όντας το τέλος μιας μακράς λίστας ε, παρατηρήσεων δεν έχω και πολλά να πω. Θα ήθελα να ε, επιστρέψω όμως σε μια βασική υποχρέωση της Ευρώπης και κυριότερα της ε, Επιτροπής για τον Πολιτισμό. Ε, φαντάζομαι ότι προτεραιότητα σε αυτήν την ψηφιοποίηση και στη δημιουργία της, ε, της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχουν τα παλιά και σπάνια βιβλία. Είναι περισσότερο ερώτηση παρά πρόταση. Θεωρώ ότι ε, ψηφιοποιώντας τα και παρέχοντας τα ελεύθερα στο διαδίκτυο προσφέρουμε πραγματικά τη δυνατότητα όχι μόνο στους νέους αλλά και στους λοιπούς Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες να χρησιμοποιήσουν βιβλία τα οποία αλλιώς βρίσκονται πολύτιμα κλεισμένα σε βιβλιοθήκες στις οποίες δεν έχει κανείς πρόσβαση. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα κέριο στοιχείο στην Ευρωπαϊάνα... θα έπρεπε να είναι ακριβώς η ψηφιοποίηση και η ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στα παλιά και σπάνια βιβλία, όπου δεν υπάρχει και το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και όπου παράλληλα προσφέρουμε μία εναλλακτική δυνατότητα συντήρησής τους. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχει γίνει κάτι τέτοιο και αν έχει το σκοπό να το περιλάβετε στο προσχέδιο για την λειτουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Ευχαριστώ. Η τελευταία παρέμβαση, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τρίπελ. Όντω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα και μεγάλου εύρου. Όλα αυτά που μα είπατε είναι πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βλέπετε, πρέπει πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε τον στόχο μας, το εύρος, γιατί καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουμε να βγούμε έξω. Η χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη περίπου. Εκτό αν θέλουμε σαν το Google κι εμεί. αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουμε. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να καθορίσουμε τι θέλουμε να το κάνουμε. Ε, αυτό που ακούσαμε είναι πάρα πολύ καλό για τους κλασικούς. Υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να καθορίσουμε ποιος είναι ο στόχο μας. Και έπειτα να δουλέψουμε σκληρά ώστε να βρούμε χρήματα. Χρηματοδότηση που από ό,τι φαίνεται και από όσα μας είπατε είναι πολύ δύσκολο. Πριν λοιπόν μπούμε στην ουσία που είναι πάρα πολύ καλή, προσοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί ήσασταν πολύ που πραγματικά δείξατε ενδιαφέρον και προτείνατε ιδέες για τη συζήτηση αυτή. Το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι πρώτον το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού, το περιεχόμενο ε, και πώς εμείς μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις γνώσεις, αυτό το περιεχόμενο καλύτερα από άλλους και δεύτερον βεβαίως και πολύ σημαντικό χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Επαναλαμβάνω, σας πρότεινα μια τελευταία ιδέα, το θέμα του προϋπολογισμού για την ε, επικοινωνία. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και τον τραπεζικό τομέα. Εγώ δεν είμαι κατά. Είτε να βρούμε χορηγούς, sponsoring. Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Όχι συγκεκριμένα η Mercedes, η Nokia, η Coca-Cola, αλλά να υπάρχει μία φράση που να λέει το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από τους εξής χορηγούς. Τελείωσε μία φορά και αυτό αρκεί. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση εν μέσω των λογοτεχνικών έργων. Επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση με την Google δεν θα είναι εύκολη. Πρόκειται για έναν τεράστιο φορέα, ο οποίος κινείται γρήγορα, είναι αποτελεσματικός και βεβαίως θα πρέπει, όπως είπε και η Χέλγα, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ όλους που πήραν το λόγο. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες ε, ιδέες. Θα πάρω το λόγο καταρχήν για να σας μιλήσω για τις γενικές κατευθύνσεις. Όσον αφορά το Google, όντως υπάρχει η εμπορική προσέγγιση αυτής της ε, ψηφιακής διάθεσης έργων. Η διάθεση από το Google έχει σίγουρα πλεονεκτήματα. Πρώτον, αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, ταχύτητα. Υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά σημεία ότι η διαχείριση της γνώσης γίνεται με έναν καθαρά εμπορικό τρόπο. Και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι δεν είναι δυνατόν η ποιότητα να μην πληγεί από αυτήν την καθαρά εμπορική διάθεση και διαχείριση. Το μοντέλο λοιπόν του Google είναι ταχύτατο, είναι αποτελεσματικό, είναι γνωστό στους νέους, είναι ενδιαφέρον λοιπόν, αλλά αυτή η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα ακολουθείται και από μια ολόκληρη ε, σειρά εκτιμάτων και αρνητικών σημείων. Η συζήτηση λοιπόν συνεχίζεται. Δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και για να μην τη χάσουμε πρέπει και εμείς να τη δράσουμε γρήγορα με πολιτικές ιδέες και με δέσμευση. Θεωρώ ότι πέρα από τη συζήτηση που θα έχουμε εδώ σαν Επιτροπή Πολιτισμού, γιατί σαφώς και πρέπει εμείς να πάρουμε θέση, θα πρέπει επιγόντως να έρθουμε σε επαφή με όλα τα Υπουργεία Πολιτισμού αλλά και τα Υπουργεία Οικονομικών των χωρών μας, γιατί αυτοί είναι που θα μας στήριξουν καταρχήν. Δεν πρέπει εμείς εδώ στην Ευρώπη αποκομμένοι και απομονωμένοι να προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκό το οποίο κανείς δεν θα ξέρει τι είναι και δεν θα ενδιαφέρει κανέναν. Πρέπει πραγματικά να έρθουμε σε επαφή άμεσα με τους υπουργούς πολιτισμού οι οποίοι θα πρέπει να προωθήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, το θέμα αυτό, να γίνει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο να γίνει γνωστό στις ευρωπαϊκές χώρες και με τους Υπουργούς Οικονομικών, γιατί χωρίς τη δική τους απόφαση δεν πρόκειται να μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Θα ξεκινήσουμε μια πολιτική, αν θέλετε, κινητικότητα, αλλά για να προχωρήσει το θέμα θα πρέπει και οι Υπουργοί Πολιτισμού στα κράτη-μέλη και οι Υπουργοί Οικονομικών να μας στηρίξουν. Εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση, όχι μόνο εδώ, αλλά και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, πολλά μοντέλα υπάρχουν. Υπάρχουν θεωρητικά μοντέλα και υπάρχουν και ρεαλιστικά μοντέλα. Μία κρατική χρηματοδότηση σε κάποιες χώρες αυτό είναι πιο εύκολο από ότι σε άλλες. Υπάρχουν ε, κρατικές βιβλιοθήκες, υπάρχει η λεγόμενη ίση πρόσβαση κοινωνική πολιτική που στηρίζει την ε, πρόσβαση όλων των νέων και των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων στη γνώση. Αυτό είναι κάτι που βεβαίως και όλοι το επιθυμούμε και στην Ευρώπη κάτι τέτοιο θα είχε πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο. Μια κρατική λοιπόν ε, χρηματοδότηση είναι ιδανική, αλλά είναι εύκολο να επιτευχθεί άμεσα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω όμως ότι η χρηματοδότηση θα έρθει πιο γρήγορα από τον προϋπολογισμό e-content. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπάρχει το κανάλι της ψηφιακής διάθεσης των έργων, στο οποίο θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να ε, ξεκινήσουμε και να βρούμε την πρώτη μας χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν από πολιτικής απόψεως να συμφωνήσουμε πού θα στραφούμε για τη χρηματοδότηση και τέλος, όποιες άλλες πηγές χρηματοδότησης προσθεθούν σε αυτή την πρώτη μας προσπάθεια είναι βεβαίως ευπρόσδεκτες. Χορηγή, sponsoring, ε, εταιρική σχέση ιδιωτικού τομέα και δημόσιου. Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι επίσης ευπρόσδεκτες. Θα πρέπει βεβαίως να εξετάσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και ιδιωτικά κονδύλια ε, πρέπει να προσελκύσουμε. Η Ντόρις είπε μόλις τώρα ότι η Ευρώπη θα πρέπει καταρχήν να διαθέσει κάποια κονδύλια και να εξηγήσουμε σε όλους όσους δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον ότι όπως ακριβώς γίνεται και στην Αμερική σε μια εποχή οικονομικής κρίσης αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι μακροπρόθεσμες. Η ψηφιακή διάθεση των έργων είναι κάτι που δεν πρέπει να το δούμε με προοπτική μηνών ή των επόμενων δύο-τριών ετών. Το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι Meet the Europeana. Συναντήστε, ελάτε να δείτε τι είναι το Europeana. Με αυτόν τον τρόπο θα προκαλέσουμε το ενδιαφέρον και βεβαίως Υπάρχει και το θέμα της διαφήμισης, πώς δηλαδή μέσω της διαφήμισης, τηλεοπτικά σποτ και άλλο είδους διαφήμιση μπορούμε επίσης να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του κοινού ε, για το ευρωπαίαν. Αυτό βεβαίως υπό όρους και προϋποθέσεις. Σε γενικές γραμμές μπορεί κανείς να πει ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι που μοιάζει με αυτό που κάνει το Google, που να μην βασίζεται όμως μόνο στην διαφήμιση. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός φορέας ρύθμισης και αυτό βεβαίως είδα ότι όλοι ε, που πήρατε το λόγο συμφωνείτε. Το θέμα τώρα των πνευματικών δικαιωμάτων, του copyright. Ναι και όχι, ναι και όχι. Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά βεβαίως θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους εγγραφείς αυτούς, οι οποίοι βεβαίως μπορούν να εγκαταλείψουν το copyright. Γιατί, διότι παραδείγματος χάρη κάποιος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, έχει ένα μισθό, οπότε δέχεται το σύγγραμμά του ή το βιβλίο του να διατεθεί δωρεάν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι οι οποίοι ζουν από τα έργα τους και για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ε, εγκαταλείψουν αυτά τα εισοδήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Εγώ είμαι κατά της πρόσκοπτης πρόσβασης, της πρόσβασης δωρεάν σε περίπτωση όπου οι δημιουργοί και οι συγγραφείς είναι αντίθετοι γιατί ζουν από αυτά τα εισοδήματα. Τώρα, πώς θα ενημερώσουμε το κοινό με έντυπο υλικό, αλλά όχι μόνο βεβαίως. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό κάποια κονδύλια, στο αποθεματικό ένα 10%, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τώρα εξετάσαμε διάφορα μοντέλα χρηματοδότησης, Πιστεύω θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και χορηγούς και εταιρικέ σχέσεις ιδιωτικού τομέα και δημόσιου και κρατική χρηματοδότηση. Αλλά προς Θεού μην καθυστερήσουμε και μην αφήσουμε τον Google να μας προσπεράσει έτσι ώστε να είναι πολύ αργά. Θα σε ευχαριστώ. Ναι, το έντυπο υλικό είναι σίγουρα ένας τρόπος να γίνει γνωστό το Ευρωπαϊκό, αλλά πιστεύω ότι η Γενική Διεύθυνση που ήταν χτες παρούσα, αλλά και άλλες γενικές διευθύνσεις μπορούν να μας στηρίξουν σε μια πρώτη φάση. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Φόλμαν, μου είπαν ότι είναι εδώ. Έχετε το λόγο, κύριε Φόλμαν. Um, Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα μας ικανοποιεί η ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, η έκθεσή σας. Και όπως είπανε πολλοί ομιλητές, είναι θεμελιώδες το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης να είναι προσβάσιμη στους πολίτες. Όπως υπογράμμισαν βέβαια πολλοί ομιλητές, θα έπρεπε εξαιτία και του Google και εξαιτία των γενικότερων συζητήσεων που γίνονται, να δούμε το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλέπετε αυτό που έγινε στην Αμερική είναι αυτό που έκαναν και την Ευρώπη να αντιδράσει. Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά υπάρχει. προσύ σε πάνω από 4 με 6 εκατομμύρια θέματα, παλιά βιβλία, μελέτες, Δοκιμάστε το. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα, στο ίντερνετ και θα δείτε ότι θα βρείτε ήδη πολλά πράγματα. Και θα καταλάβετε και τι δυνατότητες έχει το Ευρωπαϊκό παραπέρα. Ελπίζω και προσδοκώ συνεργασία με την εισηγήτρια και τους κοιόδους εισηγητές εφόσον το επιθυμούν. Και είμαστε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Περιμένουμε το σχέδιο έκθεσης και θέλουμε φυσικά να ενημερωθούμε για τις διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα βασικά. Ευχαριστούμε κύριε Φόλμαν. Βλέπω ότι και το Συμβούλιο είναι εδώ. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου λοιπόν. Του ζητάω να περάσει την ιδέα αυτή στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού και στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών. Γιατί όπως είπε και η Χέλγα, χωρίς τη δικιά τους βοήθεια τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη σημερινή συζήτηση που πιστεύω ότι βοηθάει όλες τις πλευρές. Και μπορούμε να τελειώσουμε με τη συζήτηση του θέματος αυτού. Περιμένουμε τον Επίτροπο, τον κύριο Όρμπαν. Στις 10 ήθελε να είναι παρόν. Ξέρετε ότι είναι ο Επίτροπος υπεύθυνο για την πολυγλωσία, για τη γλωσσική πολυμορφία. Θα ήθελα, συνάδελφοι, να καθίσετε, κύριε Λόκεγκαρτ. Καθίστε, παρακαλώ. Hier kommt der Lockergard hin. Ich sehe nicht ein, dass die immer unten sitzen. Du musst mich vertreten gleich. Geh nicht weg. So, jetzt zu Punkt 10 der Tagesordnung. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τον Επίτροπο, τον κύριο Όρμαν, υπεύθυνο για το θέμα της γλωσσικής πολυμορφίας. Ξέρετε ότι είναι ένα από τα σημεία κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε την μητρική μας γλώσσα, να έχουμε τα έγγραφα στη μητρική μας γλώσσα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως είναι και θα παραμείνει συνδεδεμένο σε αυτήν την αρχή ε, η μητρική γλώσσα συν δύο γλώσσες να διδάσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μια γλώσσα γειτονική της χώρας στην οποία βρισκόμαστε συν μια ευρέως διαδεδομένη γλώσσα, η lingua franca. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε που σήμερα δεχτήκατε να έρθετε να μας μιλήσετε. Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα εργασία που έχετε κάνει για το θέμα που μας απασχολεί πολύ. Τους τελευταίους μήνες είχαμε συζητήσει και ψηφίσει μια έκθεση για την γλωσσική πολυμορφία. Την πολυγλωσσία, η ήταν ο Πορτογάλος συνάδελφος Βάσκο Γκράσα Μούρα. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Πιστεύω ότι αυτά που θα μας πείτε μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, πριν από οτιδήποτε άλλο θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πακ και να τη συγχαρώ πάνω απ' όλα για τον ορισμό της στην Προεδρία της Επιτροπής μας. Συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε, λέει στα Γερμανικά ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή που μου κάνατε. Εγώ προσωπικά δίνω μεγάλη σημασία στο διαρθρωτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την δικιά σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία ε, να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις κοινέ μας δραστηριότητες και προκειμένου να δω ποιες είναι οι δικές σας αντιδράσεις απέναντι στις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, επίτροπος δηλαδή υπεύθυνο για την πολυγλωσία, έθεσα ως στόχο μου να εξετάσω τους στόχους και τα θετικά της πολιτικής μας στον πολιτιστικό τομέα, έτσι ώστε να ενισχύσω τις αρμοδιότητές μας, την κινητικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Αυτές είναι κάποιες βέβαια μόνο πτυχές της πολιτικής μας. Τώρα θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες από τις πρωτοβουλίες μας προκειμένου να αναπτύξουμε την πολιτική μας αυτή υπέρ της πολυγλωσσίας. Στη συνέχεια, κάπω σύντομα, θα αναφερθώ στα επιτεύγματά μας και τέλος θα αναφερθώ στους στόχους, της προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια. Για να δημιουργήσουμε μια φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της πολυγλωσσίας, ήταν πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο να λάβουμε υπόψη μας νέες ιδέες, απόψεις και προτάσεις από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα αναλύοντας τις συστάσεις των δύο ομάδων υψηλού επίπεδου εμπερογνωμόνων και προσωπικότητων. Πρώτα έχουμε ένα, μια ομάδα υψηλού επίπεδου για την πολυγλωσία που έκανε προτάσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την εκμάθηση όλων των ξένων γλωσσών των περιφερειακών επίσης γλωσσών, των μειονοτικών και των γλωσσών των μεταναστών. Έπειτα υπάρχει μια συμβουλευτική ανεξάρτητη ομάδα στην οποία συμμετέχουν διανοούμενοι που ονομάζεται η ομάδα Μαλούφ. Η ομάδα αυτή λοιπόν ανέλησε το ρόλο που παίζουν οι ξένες γλώσσες στην ολοκλήρωση και τον πολιτισμικό διάλογο. Επίσης προσκάλεσα τους Υπουργούς Παιδείας των κρατών μελών σε μια διάσκεψη προκειμένου να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, κοινή δέσμευση υπέρ της βελτίωσης της πολυγνωσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά έγινε συζήτηση σε υπουργικό επίπεδο και που ασχολήθηκε δηλαδή με αυτό το θέμα της πολυγλωσσίας αποκλειστικά. Άκουσα επίσης και άλλες πλευρές, όλα τα κοινοτικά όργανα, όλους τους ενδιαφερόμενους, για να δω τι μορφή θα έπρεπε να πάρει η πολιτική μας ώστε να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των πολιτών. Αυτά που εσείς προσφέρατε στο διάλογο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικά, η Επιτροπή σας δηλαδή. Δημιουργήσαμε επίσης και ένα φόρουμ επιχειρήσεων για την πολυγλωσία. Αυτό είναι ένα φόρουμ όπου συγκεντρώνονται πολλοί ειδικοί για να αναλύσουμε τον αντίκτυπο των πολιτικών μας στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τι αποτέλεσμα είχαμε τώρα από αυτήν την τόσο πλούσια εμπειρία. Τι πετύχαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2008 υιοθέτησε την ανακοίνωσή της «Πολυγλωσία, ένα πλονέκτημα για την Ευρώπη και μια κοινή δέσμευση». Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τους διάφορους τρόπους που προτείνουμε για την πρόθεση της πολυγλωσσίας και αυτό μέσα από πολλές πολιτικές είναι ένα εγκάρσιο μήνυμα. Η πολιτιστική πολυμορφία και η γλωσσική πολυμορφία είναι και το κλειδί υπέρ της ε, προσωπικής ταυτότητας του καθενός μας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι η πολυγλωσσία αποτελεί πλούτο, αποτελεί πλεονέκτημα για όλους μας. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε δηλαδή σαν ένα εμπόδιο, κάθε άλλο. Ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής μας παραμένει το στίχημα που βάλαμε για να πετύχουμε τους στόχους της Βαρκελόνης του 2002. Δηλαδή η εκμάθηση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών. Ο κάθε δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης να γνωρίζει τη μητρική του γλώσσα συν άλλες δύο. Το Συμβούλιο ε, Παιδείας λοιπόν επιβεβαίωσε τον στόχο αυτό τον Εύρο του 2008 και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μέτρα προκειμένου να προωθήσει την πολυγλωσία λαμβάνοντας υπόψη και τις γλωσσικές ανάγκες των πολιτών και των θεσμικών οργάνων. 24 Μαρτίου 2009 είχαμε το δικό σας ψήφισμα για την πολυγλωσία που μας στήριξε στην πολιτική μας διότι χαιρέτησε την πολιτική μας αυτή προώθησης εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών, πέρα από την μητρική. Ότι αυτό πρέπει να ισχύει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δηλαδή. Γιατί τώρα αυτή η Ευρώπη είναι τόσο ιδιαίτερη, γιατί έχει ακριβώς μια τεράστια πολυμορφία γλωσσών και πολιτισμών. Γιατί βλέπετε κάθε γλώσσα σημαίνει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ε, μεταφέρει μνήμες, είναι πολιτιστική και λογοτεχνική κληρονομιά και αποτελεί και μια πολύ καλή βάση για την πολιτιστική ταυτότητα. Το να σεβόμαστε την γλωσσική πολυμορφία αποτελεί βάση του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Έτσι νιώθει κανείς ότι ανήκει στην Ευρώπη. Ότι επωφελείται από την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Και αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο για να αποφύγουμε την αδιαλαξία και τις συγκρούσεις. Οι πολλές γλώσσες που μιλούνται μέσα στην Ευρώπη μπορούν να αποτελήσουν και μια γέφυρα προς άλλους ανθρώπους, προς άλλους πολιτισμούς, γιατί ακριβώς ευνοεί την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μας. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου λοιπόν για την πολυγλωσία στήριξε το στόχο μας αυτό. Συμπεριλαμβανομένης και της εκμάθησης ε, γλωσσών που μιλούνται λιγότερο, περιφερειακών γλωσσών. Είπαμε ότι οι γλώσσες αποτελούν ένα πολιτιστικό πλεονέκτημα. Πρέπει λοιπόν να τις προστατεύσουμε για να τις τροφοδοτήσουμε. Η γλωσσική πολυμορφία επίσης ευνοεί και την ευημερία. Και υπάρχει πολύ στενή σχέση ανάμεσα στην γνώση ξένων γλωσσών και τη δυνατότητα να μπορέσει κανείς να βρει δουλειά. Οι επιχειρήσεις και οι μεγάλες και οι μικρές προσπαθούν να έχουν προσωπικό που γνωρίζει ξένες γλώσσες οι γλώσσες αυτές αποτελούν ένα συν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σίγουρα τα αγγλικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο διεθνές επίπεδο για τις επιχειρήσεις, αλλά δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές ανάγκες. Πριν από λίγο, το Σεπτέμβριο, δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα για έναν συνεχή διάλογο με τις επιχειρήσεις, με τους κοινωνικούς εταίρους και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έχοντας αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές, θα καταλήξουμε σε λύσεις προκειμένου να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Κυρίως μας ενδιαφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί πολλές φορές αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αρκετούς πόρους. Εμείς όμως δεν σταματάμε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την παγκοσμιοποίηση και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας, όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και εκτός. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και ε, μας ενδιαφέρουν και οι σχέσεις μας εκτός Ευρώπης. Και γι' αυτό και διευρύνουμε τον τομέα της πολυγλωσσίας. Έχουμε υπογράψει κοινέ δηλώσεις για συνεργασία στον τομέα της πολυγλωσσίας με την Κίνα και την Ινδία. Μεγάλο επιτεύγμα αυτό. Και μάλιστα πολύ σύντομα θα συναντηθώ και πάλι με τους Κινέζους ομολόγους μας στην ε, Φραγκφούρτη, στη Γερμανία, στην έκθεση βιβλίου εκεί. Είναι σαφές ότι ο διάλογος με τέτοιες χώρες δεν είναι πάντα εύκολος, αλλά υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και εκείνοι δηλαδή, όπως και εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες των άλλων. Έρχομαι τώρα στο πρόγραμμα της Επιτροπής για τη Διαβίου Εκμάθηση 2007-2013. Αφορά όλες τις γλώσσες. Υπάρχουν και άλλα μέσα. Υπάρχει το Erasmus Mundus για παράδειγμα και το πρόγραμμα Πολιτισμός. Είναι μέσα τα οποία μας βοηθούν να μαθαίνουμε γλώσσες από τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης δηλαδή. Εμείς θέλουμε όντω να πάμε πέρα από τα προγράμματα, πέρα από τα σύνορα. Θέλουμε να αποφεληθούμε από ό,τι ευκαιρίες μπορούν να προσφερθούν για να μάθουμε ξένες γλώσσες τους Ευρωπαίους. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η πολυγλωσσία είναι ένα εγκάρσιο χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει δηλαδή όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Έρχομαι τώρα στη λογοτεχνική μετάφραση. Αυτή κάτω από οποιαδήποτε μορφή είναι πολύ βασικό στοιχείο για να δούμε ποια είναι η νοτροπία και ποιες είναι οι συνήθειες των λαών της Ευρώπης. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν των προνομίων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ε, λογοτεχνική μετάφραση. Πρόσφατα μάλιστα με τον πρόεδρο Μπαρόσο ξεκινήσαμε μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη σημασία που έχει η λογοτεχνική μετάφραση ως μέσο ολοκλήρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Επίσης, πρέπει να αναφερθώ εδώ και στην ε, διοργανική διάσταση της πολυγλωσσίας. Ξεκίνησα τη θητεία μου 1η του 2007. Ε, από τότε έχουν προσθεθεί τρεις νέες γλώσσες. Έχουμε φτάσει στις 23 γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βουλγαρικά, τα ιρλανδικά και τα ρουμανικά συμπεριλήφθηκαν με μεγάλη επιτυχία στα ευρωπαϊκά κοινωτικά όργανα. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Καταφέραμε να έχουμε ένα νέο ρεκόρ παραγωγής. Έχουμε μεταφράσει περίπου 5 εκατομμύρια σελίδες σε λιγότερο από τρία χρόνια. Αυτή είναι μια αύξηση τεράστια, η οποία όμως δεν περιόρισε τον ε, στόχο μας για ποιότητα στις μεταφράσεις, κάθε άλλο. Χρησιμοποίησαμε νέα μέσα, νέες μεθόδους, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα. Και όχι η μετάφραση αυτή να χαλάσει όσον αφορά την ποιότητά της. Κάθε άλλο. Για να διατηρήσουμε τώρα την ποιότητα αυτή, ζήτησα μάλιστα και από τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας να συγκροτήσει μία ομάδα προβληματισμού με ειδικού που ονομάζεται μάλιστα Φόρουμ Προβληματισμού για την Πολυγλωσία και την Κατάρτιση Νεοδιερμηνέων. Και αυτό για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν για νομικούς διερμηνείς και πώς μπορεί η κατάρτιση αυτή να βελτιωθεί. Στις αρχές λοιπόν του 2009 το φόρουμ αυτό υπέβαλε έκθεση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει συστάσεις για ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα ευρωπαϊκό στον τομέα της ε, ε, διερμηνίας για νομικούς. Θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο οδηγίας πάνω σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη στα κοινωτικά όργανα από αυτή στην οποία μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάντως, ο στόχος μας είναι ο εξής. Να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα, μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν αυξηθεί ο αριθμός των επίσημων γλωσσών. Ο στόχος όμως αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον βελτιωθεί η τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας και εφόσον βέβαια έχουμε και περισσότερους πόρους για τις γλωσσικές υπηρεσίες των κοινωτικών οργάνων. Πρέπει να βρούμε τους καλύτερους για να συντονίσουμε επίσης τη ζήτηση, να τη συντονίσουμε με τη τεχνολογία που διαθέτουμε. Και σε αυτό μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να βοηθήσουν. Έχουμε κάνει πολλά βήματα προς τα μπρος για να προωθήσουμε την πολυγλωσία. Μένουν όμως να γίνουν ακόμα πολλά τα επόμενα χρόνια. Από την αρχή υπογραμμίσαμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Γιατί θέλουμε να σεβόμαστε την επικουρικότητα. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι στόχοι μας είναι στόχοι κοινοί με εκείνους των κρατών μελών. Επίσης, μας ενδιαφέρει ο διαρθρωμένος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πολιτική μας πρόθεση της πολυγλωσσίας. Σύντομα θα ξεκινήσουμε ένα φόρουμ με όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, της μη επίσημης εκπαίδευσης, για να βελτιώσουμε την προσέγγιση στην πολυγλωσία για να βελτιώσουμε μάλλον την πρόσβαση στην πολυγλωσία εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν κοντά σε αυτήν. Υπάρχουν πολλές ιδέες. Τώρα, πιστεύουμε ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών πρέπει να γίνεται πολύ νωρίς. Σε νεαρή ηλικία δηλαδή. Είναι προφανές από ό,τι φαίνεται ότι όσο πιο νωρίς μάθει κανείς ξένες γλώσσες, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχει να κερδίσει σε προσωπικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης για τους γονείς πάνω απ' όλα. Πρόκειται για μια εκστρατεία η οποία στηρίζει και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι τώρα στη στήριξη των γλωσσών των μεταναστών. Το 2008 είπαμε ότι οι μετανάστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν την ε, γλώσσα της χώρας στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Αυτό τους βοηθάει να νιώθουν καλύτερα ότι ανήκουν στην κοινωνία εκείνη μέσα στην οποία ζουν, ε, προστατεύει την αξιοπρέπειά τους, και σίγουρα βοηθάει το διαπολιτισμικό διάλογο. Όμω πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά. Εμεί πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να δείξουν ότι σέβονται και τις γλώσσες, τις μητρικές γλώσσες των μεταναστών που έχουμε. Άρα πρέπει να βρούνε τρόπους για να χρησιμοποιούν αυτές τις γλώσσες μέσα στις επιχειρήσεις. Αυτό γιατί πιστεύουμε ότι οι γλώσσες τρίτων χωρών μπορούν να είναι χρήσιμες για να ενισχυθεί η οικονομική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Τα γενικά θέματα εκμάθησης γλωσσών από πλευρά των μεταναστών είναι θέμα που αποτέλεσε στρατηγικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το στόχο του 2020. Πρόκειται πάνω απ' όλα για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας στην οποία ζουν οι μετανάστες, που προέρχονται δηλαδή από άλλες χώρες, αλλά όπως σας είπα μας ενδιαφέρει και η εκμάθηση της γλώσσας των μεταναστών από τους άλλους Ευρωπαίους. Το πρόγραμμα διαβίου κατάρτισης έχει συνεισφέρει στην προώθηση της εκμάθησης γλωσσών. Τώρα πρέπει να δούμε το νέο πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το 2014, πώς αυτό λοιπόν θα ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και πώς θα μας βοηθήσει να έχουμε περισσότερο γνώσεις για άλλους πολιτισμούς, για άλλες συνήθειες και πώς θα βοηθήσει και την κινητικότητα. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Μπαρόσο μας πρότεινε μία πρωτοβουλία που ονομάζεται «Η νεότητα σε κίνηση». Είναι ένα είδος έρασμος για όλους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει σε όλους τους νέους να μπορούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό κάποια στιγμή. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία ενίσχυσης των γλωσσικών γνώσεων σε όλη την Ευρώπη. Το 2011 από την άλλη μεριά θα λάβει η χώρα μία διπουργική διάσκεψη προκειμένου να αξιολογήσει τους στόχους της Βαρκελόνης. Στη διάσκεψη αυτή θα ξαναδούμε τις πολιτικές μας όσον αφορά την πολυγλωσία. Και πώς θα αλλάξουμε, πρέπει να αλλάξουμε κάτι από το 2012 και μετά. Εννοείται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε προχωρήσει πολύ. Ξεκινήσαμε με ένα λευκό χαρτί ξεκινήσαμε με προσπάθειες ατομικές. Όμως μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ένα ρεύμα υπέρ της πολυγλωσσίας. Πολλοί βοήθησαν σε αυτό. Όπως σας είπα και πριν, όμως μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Είμαι πεπισμένος ότι η πολιτική αυτή αξίζει κάθε προσπάθεια. Και αυτό το διαπιστώνω και καθημερινά σε όλες τις επισκέψεις που έχω κάνει μέχρι τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη για να προωθήσω την πολυγλωσία. Διαπιστώνω καθημερινά το ενδιαφέρον των πολιτών για την πολιτική μας. Και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται και προκειμένου η πολυγλωσία να εφαρμόζεται εγκάρσια, σε όλες δηλαδή τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαι πεπισμένος ότι και εσείς συμφωνείτε μαζί μου, εσείς που βρίσκεστε τόσο κοντά στους πολίτες, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο στόχος μας είναι μεγάλος. Χρειάζεται διάλογος, διαπολιτισμικός διάλογος, θέλουμε ευημερία, ένταξη στις κοινωνίες μας στο μέλλον θα χρειαστούμε περισσότερα χρήματα. Και πάνω απ' όλα θα χρειαστούμε καινοτόμε λύσεις. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την ε, γλωσσική μας λειτουργία σε εσωτερικό επίπεδο. Με τη στήριξή σας λοιπόν, μια που εσείς είσαστε νομοθετικό και δημοσιονομικό σώμα, θα μας στηρίξετε έτσι η πολυγλωσία θα συνεχίσει το δρόμο της. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τώρα τα σχόλιά σας. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar, für die Darstellung Ihrer Politik, was Sie... Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για αυτή την δήλωση, για τα όσα κάνετε και τα τι σκοπεύετε να κάνετε. Φαντάζομαι ότι από την παρουσίασή σας θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πολυγλωσία συνδέεται περισσότερο με όλο και περισσότερο μάλλον με τις οικονομικές δυνατότητες. Είπατε πως τα αγγλικά είναι απαραίτητα ώστε να μπορεί κανείς να γίνει κατανοητός διεθνώς αλλά και στον εμπορικό κόσμο, αλλά δεν αρκεί. Γι' αυτό και θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν περισσότερες γλώσσες. Επίσης αναφέρατε πόσο σημαντικό είναι το να γίνει η ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών ώστε να μπορούν να μαθαίνουν τη δική τους μητρική γλώσσα αλλά να μπορούν ταυτόχρονα να μαθαίνουν και την γλώσσα της χώρας υποδοχής διότι διαρκώς βρίσκονται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημαντικά θέματα τα οποία αγγίξατε και έχω εδώ έναν μακρύ κατάλογο ομιλητών. Πρώτα ο κύριος Τσβέρ. E, najprej bi se vam rad zahvalil za zelo celovito sliko e, predstavitev vašega dela. Na... Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν Επίτροπε για την πολύ ωραία σας παρουσίαση και την πολύ κατανοητή σας παρουσίαση. Ε, πριν από τρία χρόνια, η Επιτροπή, νομίζω περίπου τρία χρόνια ήταν, ε, προσπάθησε να θεσπίσει μια συγκεκριμένη εντολή και φυσικά να προωθήσει έτσι την πολυγλωσία. Και θα πρέπει από αυτού να σας συγχαρώ. Ίσως τα επόμενα χρόνια η Κομισιόν να μπορούσε να φτιάξει μια, κάποιους δείκτες γλωσσών ώστε να δούμε τις γλωσσικές δεξιότητες στην Ευρώπη και να κάνουμε και συγκρίσεις. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει αρχικά σε πιλωτικό στάδιο και σε συνδυασμό με την ε, Επιτροπή Παιδείας. Θα μπορούσαμε να δούμε λοιπόν πώς προχωρούν οι γλώσσες, αλλά φυσικά το καλύτερο θα ήταν να ληφθούν υπόψη όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες και φυσικά αυτό συνδέεται με τους ε, οικονομικούς πόρους, τα κονδύλια, αλλά θα ήμασταν υπέρ του να προωθηθούν όχι μόνο οι επίσημες γλώσσες, αλλά και οι γλώσσες των γειτονικών μας χωρών αλλά και χώρες, οι γλώσσες με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι Ευρωπαίοι. Ίσως θα θυμάστε και ήδη αναφέρθηκε πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνει κανείς την γλώσσα του γειτονά του. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να μιλά τη γλώσσα κάποιας ε, εθνιωτικής ομάδας, όταν ας πούμε έχεις ε, κάποιες ε, μειονότητες στη χώρα σου και ιδιαίτερα σημαντικό είναι βέβαια για τους νέους της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίσας. Α. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πληρέστατη. Η πολυγλωσία είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει εμένα όλος ιδιαίτερος. Ίσως επειδή η πολιτική μου διαδρομή να είναι ατυπική. Είμαι και Ισπανός και Καταλανός και ήμουν και υπουργό Πολιτισμού για χρόνια στην Ισπανία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκμάθηση ξένων γλωσσών και αναγκαία. Ξέροντας από την εμπειρία που έχω εγώ ε, στη Μαδρίτη που έχουμε σχολεία ε, ισπανικά, αγγλικά και γαλλικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για τους νέους. Συμφωνώ όμω, και με αυτά που είπε και ο συνάδελφος πριν, ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε στην εκμάθηση των πιο συνηθισμένων γλωσσών ή των πιο σημαντικών. Είναι εξίσου ενδιαφέρον να μαθαίνουμε και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Εσείς αναφερθήκατε στη στήριξη της γλώσσας των μεταναστών. Είναι θετικό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πριν στηρίξουμε τη γλώσσα των μεταναστών ότι θα υπάρχει στήριξη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχουμε τέσσερις επίσημες γλώσσες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο τα ισπανικά. Τα καταλανικά, πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι τα μιλάμε, και τα Βασκικά και τα γκαγέγο. Όλες αυτές είναι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεν σε διάφορα έγγραφα, αλλά δεν έχουμε ας πούμε διερμηνία. Έπειτα υπάρχει και το πρόβλημα των μειονοτικών γλωσσών, όπως τις λέμε, που ομιλούνται σε τρίτες χώρες και που άπαξ και είναι, ε, τα, είναι μια επίσημη γλώσσα, όπως είναι με τα ουγγρικά και τα σλοβακικά στις δύο αυτές χώρες, δημιουργούνται προβλήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μένα η γλώσσα δεν είναι θέμα κράτους, είναι θέμα ανθρώπων και άρα πρέπει να σεβόμαστε τη γλώσσα του καθενός των ανθρώπων. Και στην περίπτωση των μεταναστών ναι, αλλά πριν φτάσουμε στους μετανάστες ας βάλουμε λίγη τάξη στα δικά μας, στις δικές μας γλώσσες δηλαδή τις ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Χάνιμπορτ. Σας ευχαριστώ. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Είμαι Αγγλίδα, Αγγλόφωνη. Και πραγματικά είναι τεράστιο το πρόβλημα των γλωσσών. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που προτείνατε, να γίνει ένα είδος αξιολόγησης ε, της ε, εκμάθησης των γλωσσών. Σε εμά στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε καθηγητές που να διδάσκουν σωστά τις ξένες γλώσσες, γιατί ίσως δεν υπάρχει αρκετή ανάγκη. Αυτό βεβαίω είναι αντίθετο με όλα όσα λέμε εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω μεταξύ άλλων. Τι είναι η πολιτική των ε, κρατών μελών. Γιατί τελικά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών του εκπαιδευτικού του συστήματος. Και αναρωτιέμαι τι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Για τις μεγάλες γλώσσες τώρα βεβαίως αναφέρομαι. Συμφωνώ απολύτως όσον αφορά αυτό που λέτε για τις γλώσσες των μεταναστών. Έχω προσωπική εμπειρία. Εξάλλου είμαι και στο Συμβούλιο το Διοικητικό ενός σχολείου στο Λονδίνο με 39 διαφορετικές γλώσσες. Βεβαίως και οι μετανάστες πρέπει να μιλούν την γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και την μητρική τους γλώσσα. Και είναι πολύ σημαντικό για την ενσωμάτωσή τους να μπορέσουν να κρατήσουν και τη μητρική τους γλώσσα. Και θα ήθελα να μάθω τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό πάντως να αναγνωρίσουμε την γλώσσα των μεταναστών. Άκουσα επίσης και τον Ισπανό συνάδελφο, που μιλάει για τις μειονοτικές γλώσσες στο εσωτερικό μιας χώρας. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι οι γλώσσες όπως τα ουαλικά, παραδείγματος χάρη, τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε, θα πρέπει να τα στηρίξουμε. Δηλαδή, κοινότητες στο εσωτερικό μιας χώρας που μιλούν μια γλώσσα μειονοτικοί, θα πρέπει κάπως να τους στηρίξουμε και να μπορέσουν να συνεχίσουν ε, να μιλούν τη γλώσσα τους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Τούκες έχει Elnök asszony, biztos úr, stimát komisszár, tisztelt biztos úr, romániai magyarként. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι Ούγγρος από τη Ρουμανία. Και καταλαβαίνετε ότι με ενδιαφέρει διπλά το θέμα το οποίο αναφέρατε. Σας συγχαίρω κύριε Επίτροπε, καθότι οι προσπάθειες που κάνετε είναι πραγματικά άξιες να υποστηριχθούν από όλους μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα γιατί μεταξύ άλλων είπατε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε γλώσσες οι οποίες δεν είναι οι γνώσεις της πλειοψηφίας σε μια χώρα, όπως τώρα, τα σκοτσέζικα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά την χρήση των γλωσσών, έχουμε τρεις κατηγορίες, αν θέλετε, γλωσσών. Έχουμε τους υποψήφιους, έχουμε τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε βεβαίως και τις τρίτες χώρες. Αυτές οι τρίτες χώρες τις οποίες εξάλλου και αναφέρατε στην παρουσίασή σας όταν μιλήσατε για τις άλλες γλώσσες. Σε μια άλλη επιτροπή στην οποία είμαι μέλος μιλήσαμε ακριβώς για αυτό το θέμα, τις γλώσσες αυτές οι οποίες απειλούνται. Ξέρετε παραδείγματο χάρη ότι υπάρχουν διακρίσεις στην Κίνα παραδείγματο χάρη και στην Κίνα υπάρχουν πολλές γλώσσες οι οποίες δεν είναι γλώσσες που ομιλούνται από ένα μεγάλο αριθμό πολιτών. Στην Σερβία επίσης, στην Ουκρανία παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Και βλέπουμε ότι τα Ούγγρικα είτε τα Ρουμάνικα είναι θύματα διακρίσεων στην Ουκρανία, παραδείγματο χάρη. Μπορεί κανείς να πει ότι η χρήση των μειονοτικών γλωσσών, όπως τα ουγγρικά ή τα, τα ρουμάνικα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουν. Ζητώ λοιπόν εδώ από την Επιτροπή να προσέξει ιδιαίτερα τι γίνεται στις χώρες αυτές. Στη Σερβία τα ρουμάνικα που ομιλούνται από τη ρουμανική μειονότητα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και καταλαβαίνετε ότι μέσω της γλώσσας περνάει και η ταυτότητα αυτών των Ρουμάνων. Στη Μολδαβία επίσης. Ο Πρωθυπουργός ε, της ε, Δημοκρατίας του Μόλδοβα Μα είπε ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει πλέον γλώσσα που να χαρακτηρίζεται σαν γλώσσα των Μολδάβων και η επίσημη γλώσσα είναι πλέον τα Ρουμάνικα. Έτσι έχουν αποφασίσει. Όσον αφορά τώρα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, Σλοβακία. Υπάρχει ένας απαράδεκτος νόμος για τις γλώσσες. Πρόκειται για ένα φασιστικό νόμο, ο οποίος υιοθετήθηκε στη δεκαετία του 30, εποχή που εμπνεύστηκε μάλιστα από τον Φράνκο, ήταν η πολιτική τότε για την εξάλληψη των μειοτήτων. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα καθεστώς τύπου Βυσσή ή ένα καθεστώς το οποίο πραγματικά δεν αρμόζει σε μια χώρα η οποία ε, θέλει να λέγεται χώρα των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τη Μακεδονία. Οι Μακεδόνες επίσης έχουν πρόβλημα γλωσσικό. Ζητώ λοιπόν από εσάς κύριε Επίτροπε, πέρα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ιδέες και τα ιδεώδη, να συγκεντρωθούμε και να προσέξουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη τα πανεπιστήμια τα ογκρικά στη Ρουμανία, η απαγόρευση της χρήσης των γλωσσών κάποιων μειονοτήτων πολύ συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah, thank you, Mr. Um, to touch a Επίτροπε Ορμπάν, θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση σε σχέση με τα όσα είπε ο κ. Τούκες τώρα. Στην ομιλία σας μη... είπατε για πολυγλωσία και για Κίνα και Ινδία. Γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω όταν συνομιλείτε με τις Κινέζικες Αρχές για το θέμα της πολυγλωσίας. Ξέρω πως πολλοί οι Κινέζοι φοιτητέ αυτή τη στιγμή μαθαίνουν ευρωπαϊκές γλώσσες και ορισμένες φορές είναι πραγματικά εξαιρετικοί στην εκμάθηση των ευρωπαϊκών γλώσσων. Το άλλο όμως που γνωρίζουμε είναι ένα πολυεθνικό κράτος. Ξέρουμε ότι οι Θηβετιανοί και εσείς αναφέρατε και το Τσιν Γιάνγκ, ε, είπατε ότι εκεί ε, δεν είναι τόσο εύκολο να μιλούν τη γλώσσα τους, να εκπαιδεύονται στην γλώσσα τους ε, στα Θηβετιανά ή την, τουρκική τουρκικής οικογένειας γλώσσα ε, στο Ήγο, αλλά θέλω να ξέρω αν όταν το συναντάτε θίγεται αυτό το πρόβλημα της πολυγλωσσίας εντός της Κίνας. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Στάκουλα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ορμπάν για την εξαιρετική εργασία που έκανε στον τομέα της πολυγλωσίας. Η παρουσίασή του ήταν εξαιρετική και μπορώ να πω μόνο ότι η γλώσσα αποτελεί την βάση της ταυτότητας. Και αν θέλουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη των πολιτών, που όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τότε το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο του οποίου η γλώσσα αποτελεί ένα ε, αναπόσπαστο τμήμα, είναι πολύ σημαντικό και μέσω των γλωσσών μπορούμε πραγματικά να μάθουμε, να γνωρίσουμε καλύτερα αλλήλους. Η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι κάτι επί το οποίο οικοδομούνται όλα τα υπόλοιπα. Οι εσωτερικές, εξωτερικές πολιτικές, πολιτική ασφάλεια και ούτω καθεξής. Εγώ έχω μια ερώτηση, σχόλιο που έχει να κάνει με τις μειονότητες. Το συζητάμε αυτό στην Ένωση ε, εδώ και πολύ καιρό. Και ελπίζω πως το θέμα αυτό θα προωθηθεί και κατά τη διάρκεια της επόμενης ε, θητείας της Επιτροπής. Όσον αφορά λοιπόν τους αυτόχθονες, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να, μάθουν, να μαθαίνουν τις γλώσσες τους, γιατί το, μέτρο του πολιτισμού μας είναι το πώς ε, αντιμετωπίζουμε τις μειονότητες. Και είμαστε τόσο δυνατοί όσο είναι η πιο αδύναμή μας, ε, ο πιο αδύναμος μας πολιτισμός. Για παράδειγμα, Στη Φιλανδία το θέμα το γλωσσικό των Σάμι στη Λαπωνία είναι εξαιρετικά σημαντικό και αν έχουμε πόρους, τους πόρους έρχονται και ακόμα και εκτός από την Ευρώπη. Υπάρχουν ε, μειονότητες στη Ρωσία. Και η πολιτική που ασκείται προς αυτές τις μειονότητες είναι αρκετά σκληρή. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να ενεργήσουμε σε ευρύτερο πλαίσιο και να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τη γλώσσα τους. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου που και πάλι να σας συγχαρώ για τόσο έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Είναι, βρισκόμαστε στη σωστή πορεία και ελπίζω πως τα πράγματα θα προχωρήσουν, θα προοδεύσουν και στην επόμενη θητεία της Επιτροπής. Η πολυγλωσία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ταυτότητάς της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάκουλα, κυρία Νέβη Νταλόβωνα και κατόπιν υπάρχουν η κυρία Κέλλη, η κυρία Παρατέλη, αλλά πρώτα πρέπει να κρατήσουμε τη σειρά. Ευχαριστώ πολύ. všetkým chválam, ktoré boli na vašu hlavu znesené. Ďakujem veľmi pekne za správu, ktorú ste nám predložili. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία που γίνεται στον τομέα αυτό και χαίρομαι γιατί έρχομαι από μια χώρα μικρή και μπορώ παρόλα αυτά να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Μιλήσατε για τους μετανάστες, μιλήσατε για τις τρίτες χώρες και τη στήριξη των γλωσσών τους. Θα ήθελα να μου πείτε πώς θα το κάνετε αυτό. Θέλετε να τους ε, χρηματοδοτήσετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θέλετε να διαθέσετε κονδύλια. Και όταν μιλάμε για πολυγλωσία και γλωσσική πολυμορφία, σε σχέση με την Κίνα, παραδείγματος χάρη, πώς αυτή η πολιτική θα μπορέσει να υλοποιηθεί εκεί. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος Τόκες στο νόμο της Σλοβακίας σας ζητώ να το διαβάσετε αυτό το νόμο. Μπορώ να σας το δώσω αν θέλετε το κείμενο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστά αυτά που είπε. Πραγματικά είναι δική του ερμηνεία αυτή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Νομίζω πραγματικά ότι είναι ακραίες αυτές οι θέσεις που ακούστηκαν εδώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ και συγχαίρω τον Επίτροπο Όρμαν για την παρουσίασή του. Αναφερθήκατε στα Ιρλανδικά, που δεν είναι επίσημη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά στην χώρα μας υπάρχει μεγάλη υποστήριξη. Ήταν σε παρακμή αυτή η γλώσσα, αλλά η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά την έκανε πιο δημοφιλή και την ε, στήριξε. ιδιαίτερα σε περιοχές ε, εκτός των πόλεων όπου ομιλείται ευρέως. Η πρωτοβουλία ε, του Προέδρου Μπαρόζο επίσης είναι εξαιρετική. Οι νέοι εν κινήσει, Youth in Move, είναι εξαιρετικά σημαντική για την εκμάθηση άλλων γλωσσών και γειτονικών χωρών αλλά και ε, άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παγιαδέλη. Thank you, Mrs. Chairman. Chairwoman. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Όρμπαν για όσα μας είπε για την πολυγλωσσία. Ε, θα ήθελα να το ρωτήσω όμως αν σκεφτήκατε ότι είναι ενδεχόμενο η, η, η ανάγκη για την διεύρυνση των γλωσσικών δυνατοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα ζητήματα από αυτά που προσπαθεί να λύσει. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Φέρχεφν, τον συνάδελφο, να μιλάει για το ιδίωμα, για, τη διά, για, για, για το ιδίωμα που μιλούν στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ε, θεωρώντας την γλώσσα. Ε, σας δηλώνω με την ιδιότητά μου την επιστημονική ότι πρόκειται για μια βουλγαρική διάλεκτο Πώς ορίζουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την γλώσσα και πώς την ξεχωρίζουμε από μία διάλεκτο. Ευχαριστώ. Okay. I I had to Ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να σας εγκαταλείψω γιατί ίσα ίσα ήταν μια ψηφοφορία που ασχολείται με τη γλώσσα της χώρας που αναφέρεται, της Μακεδονίας. Λέτε ότι είναι διάλεκτος. Αλλά είναι το ίδιο με το Λουξεμβούργο. Είναι μία διάλεκτος των Γερμανικών, είναι όμως η γλώσσα του Λουξεμβούργου. Μην είμαστε λοιπόν τόσο πολύ περίπλοκοι. Η Επιτροπή θα μας δώσει τις σωστές απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να απαντήσετε και ότι υπάρχουν σήμερα εθνικά κοινοβούλια για τα οποία προκαλούν δυσκολίες αυτού του είδους τα θέματα. Κάντε ό,τι μπορείτε για να μην τους στενοχωρήσετε. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Σβέρ. Διότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Μιλήσατε για γλωσσικούς δείκτες Είμαστε σε ένα στάδιο αρκετά προηγμένο. Το 2010 λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του δίκτυα αυτού και το 2011 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Επίσης γνωρίζετε ότι για ρεαλιστικούς λόγους, για λόγους κόστους, έχουμε ήδη ξεκινήσει με την αξιολόγηση του δίκτυα αυτού όσον αφορά τους νέους 16 ετών. Και αυτό για πέντε γλώσσες προς το παρόν. Στόχος μας όμως είναι να επεκτείνουμε περισσότερο την αξιολόγηση αυτή και να συμπεριλάβουμε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό, διότι Ακόμα και για να αξιολογήσουμε αυτές τις πέντε πρώτες γλώσσες με τις οποίες έχουμε ξεκινήσει, έχουμε δυσκολίες πέρα από τις όποιες πολιτικές ευαισθησίες που υπάρχουν και υπάρχουν. Ακόμα και για κάτι που μπορεί να φαίνεται καθαρά τεχνικό στην αρχή. Αλλά τελικά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευαισθησίες ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Γιατί να υπάρχουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο θέμα που είναι καθαρά η αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων. Και όμως υπάρχουν. Αλλά αν σκεφτούμε τώρα τον δίκτυ της πίσης, σκεφτόμαστε γιατί να είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα. Τέλος πάντων, πέρα από αυτές τις δυσκολίες όμως, υπάρχουν και άλλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα ορισμένε χώρες να μην θελήσουν να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο στάδιο του προγράμματός μας. Ελπίζουμε βέβαια τελικά να καταφέρουμε να έχουμε συμμετοχή από όλες τις χώρες μέλη και να έχουμε επίσης και αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε την αξιολόγηση αυτή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που άκουσα ότι στηρίζεται γενικά την εκμάθηση ξενογλωσσών συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσών των ε, χωρών που γυτνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και στη στρατηγική του 2005 αλλά και στη συνέχεια του 2008. Ε, είπα ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι κάτι το οποίο ενισχύει το διαπολιτισμικό διάλογο. Πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από όλες τις εντάσεις, από όλες τις συγκρούσεις, μα μόνο μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, μόνο εφόσον μπορούμε να συναντηθούμε με τα γειτονά μας, εφόσον μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του και να τον καταλάβουμε έτσι καλύτερα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης για τις συγκρούσεις και τις εντάσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για δύο κοινότητες που μιλάνε μία δίπλα στην άλλη, αν μιλάμε για μειονοτικούς πληθυσμούς που έχουμε σε ορισμένες περιοχές ή που αλλού είναι πιο πολλοί, αν μιλάμε για γείτονες χώρες, δεν έχει σημασία. Το πρόβλημα είναι πάντα το ίδιο. Μιλάμε για την ε, γνώση της γλώσσας του άλλου, έτσι ώστε να μπορούμε να τον καταλάβουμε και να συνονιθούμε μαζί του. Αυτό βοηθάει στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο κύριος Ατσβέλα τώρα, και συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά το όνομά σας, αναφερθήκατε στις ε, γλώσσες που μιλούνται στην Ισπανία. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου του 2007 ανάμεσα στα κοινοτικά όργανα και την Ισπανική κυβέρνηση άρχισε να ισχύει μια συμφωνία η οποία επιτρέπει επιπλέον διευκολύνσεις για τους Ισπανούς πολίτες, αλλά και εκτός Ισπανίας, για πολίτες δηλαδή, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις επίσημες ισπανικές γλώσσες, δηλαδή τα καταλανικά, τα βάσκικα και τα γαγέγο, τη γλώσσα της Γαλλικίας δηλαδή. Βάσει αυτής της συμφωνίας και μπορώ να σας δώσω εδώ ένα παράδειγμα, εκπρόσωποι Ισπανοί στο Συμβούλιο μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γλώσσες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πριν από λίγο, εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τα ουαλικά βάσει της συμφωνίας του 2008. Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες εκτός από αυτές. Έτσι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσαμε να αναπτύξουμε στη Βαρκελόνη ε, και να έχουμε μια ολόκληρη σελίδα στα καταλανικά με πληροφορίες για τις κοινοτικές γλώσσες, με πληροφορίες για την εκμάθηση γλωσσών κλπ. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα, πρόκειται για ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διατίθεται στα καταλανικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε όλες αυτές τις γλώσσες στα κοινοτικά όργανα και να ζητήσουν ό,τι θέλουν. Έχουν επίσης το δικαίωμα την απάντηση που θα πάρουν από τα κοινοτικά όργανα να την πάρουν στη γλώσσα στην οποία απευθύνθηκαν. Δηλαδή και στις γλώσσες αυτές που αναφέρεται. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό στις προσπάθειες που κάνουμε. Είναι προσπάθειες που κάνουμε ακριβώς για τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη. Υπάρχει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα εδώ να το υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, γιατί ίσως να μην το είπα πολύ καλά στην αρχή. Οι στρατηγικές που εφαρμόζουμε, η πολιτική πολυγνωσίας, πολυγλωσσίας που έχουμε και εφαρμόζουμε, έχουν να κάνουν με όλη τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίε μας δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνε ακόμα πιο πέρα. Συμπεριλαμβάνουν πάνω από 60 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Βέβαια, στα μέτρα του δυνατού συμπεριλαμβάνουμε και τις γλώσσες, τις μητρικές των ε, μεταναστών που έχουμε στην Ευρώπη. Τώρα θέλω να απαντήσω στην κυρία Χάνιμπολ. Δώσαμε πολύ προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στο Ηνωμένο Παρόλο που αρχικά Υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις. Στον τύπο τι διαβάζαμε. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ότι η πολυγλωσία δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία εκεί. Δεν πρέπει να είναι κάτι στο οποίο να πρέπει να επικεντρωθούμε πλήρως, μερικός μόνο. Τέλο πάντων, εμεί προσέξαμε όλου ιδιαίτερα στην κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μελετήσαμε πώ έχουν τα πράγματα εκεί. το ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα Βρετανοί πολίτες, δεν γνωρίζουν καμία ξένη γλώσσα. Εκτός από αυτό, δεν υπάρχει και κίνητρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε σαν επιχείρημα για να πείσουμε τους νέους και τους γονείς τους να καθίσουν και να μάθουν ξένες γλώσσες. Κάναμε πολλές προσπάθειες. Πολλές φορές μάλιστα μας κατηγόρησαν γιατί είπαν ότι είναι θέμα επικουρικότητας. Οπότε τι ανακατεύεστε, ότι είναι οι εθνικές αρχές, οι περιφερειακές που πρέπει να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Διαπιστώνω όμως με ικανοποίηση ότι τη σήμερα ημέρα αυτό το θέμα είναι στην επικυρότητα. Το συζητάνε και οι Βρετανικές αρχές και ο τύπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από δύο εβδομάδες, το περιοδικό The Economist δημοσίευσε ένα άρθρο που μιλούσε για τα μειονεκτήματα απέναντι στα οποία βρίσκεται ο Άγγλο πολίτη που δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα, ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Και γι' αυτό και χαιρετίζω την απόφαση που πάρθηκε από του χρόνου η εκμάθηση ξένων γλωσσών να είναι υποχρεωτική ήδη από το δημοτικό. Αυτό σίγουρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα επιφέρει αλλαγές. Από την άλλη τώρα, μετά από τις διάφορες επισκέψεις που έκανα στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώνω ότι η εμπειρία από την πολυγλωσία είναι κάτι θετικό, πολύ θετικό εκεί. Έτσι το εισπράττουν. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ πήγα σε σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πήγα σε ένα σχολείο όπου είχαν παιδιά από 100 διαφορετικές γλώσσες. 100. Τα μοντέλα ένταξης λοιπόν είναι πολύ ιδιαίτερα. Και ίσως θα μπορούσαν να εμπνευστούν από αυτά και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Ε, αναφερθήκατε επίσης στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Έχουμε το πρόγραμμά μας για την διαβίου κατάρτιση. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν υπάρχει ένα κεφάλαιο ειδικό για την πρόθεση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κεφάλαιο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη των μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών. Έχουμε χρηματοδοτήσει, για παράδειγμα, δίκτυα, το δίκτυο Cardiff, για να στηρίξουμε τέτοιες γλώσσες. Έχουμε στηρίξει επίσης και ειδικά προγράμματα για ορισμένες ε, μειονοτικές γλώσσες. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά αποτελούν μια πολύ δική στήριξη και είναι κάτι που αναγνωρίζεται από όλους όσους δουλεύουν σε αυτό το τομέα. Και συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Πριν από την αξιολόγηση που θα γίνει, νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε περισσότερους πόρους για τέτοιου είδους πολιτικές. Στον κύριο Τόκες τώρα να απαντήσω. Γνωρίζετε πολύ καλά τα περιθώρια που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οποιαδήποτε δράση της για τρίτες χώρες. Είτε είναι στην Ευρώπη είτε όχι. Εσείς αναφερθήκατε στην Ουκρανία κάποια στιγμή. Και πρέπει εδώ να σας πω ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και γενικότερα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά είναι θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμπεριλαμβάνονται σε όλες μας τις πολιτικές. Και εδώ θέλω να αναφερθώ όχι μόνο στην πολιτική γυτνίασης, αλλά μιλάω και για την εταιρική σχέση που έχουμε με τις ανατολικές χώρες. Αυτή η πολιτική είναι μια προϋπόθεση. προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη Μολδαβία. Θα ήθελα εδώ να σας πω ένα πράγμα μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις αποφάσεις των αρχών των αρχών της χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά, όταν υπάρχουν ειδικά ε, θέματα που αφορούν τα κράτη-μέλη, Αυτά τα θέματα, αυτά τα συμφέροντα μπαίνουν στο γενικό πλαίσιο και λαμβάνονται υπόψη. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο στις σχέσεις Ρουμανίας-Μολδαβίας, έχει να κάνει και στο άλλο στο οποίο αναφερθήκατε, στην τέος Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και έχει να κάνει και με τις σχέσεις της χώρας αυτής με την Ελλάδα και με τη Βουλγαρία. Και επειδή με ρωτήσατε και κάτι άλλο για την αλλαγή του γλωσσικού νόμου στη Σλοβακία. Αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος τροποποιήθηκε πριν από λίγο, πρόσφατα, από το Κοινοβούλιο και άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου του 2009. Είπα ξεκάθαρα ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη μια είμαστε υποχρεωμένοι να δράσουμε βάσει των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η γλωσσική πολιτική είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με εθνικές και περιφερειακές αρμοδιότητες. Πρέπει να σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας όταν πρόκειται για τα γλωσσικά ζητήματα. Από την άλλη βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλύει την ομοθεσία και να βλέπει αν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα η Επιτροπή αναλύει τις διατάξεις του γλωσσικού νόμου αυτού στη Σλοβακία. Και εξετάζουμε τις διατάξεις αυτές όχι μόνο για να δούμε κατά πόσο είναι συμβατές με την οδηγία 43 του 2000, που είναι οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλά επιπλέον Κοιτάμε και άλλα κοινοτικά έγγραφα, τι ισχύει δηλαδή στην εσωτερική αγορά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρίνουμε τις διατάξεις αυτές επίσης με την νομοθεσία μας για τα οπτικουστικά, για τις ετικέτες στα προϊόντα. Η ανάλυση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια ανάλυση που παίρνει χρόνο γιατί είναι περίπλοκη. Όταν όμως έρθει η στιγμή θα σας ενημερώσουμε για τα συμπεράσματά μας. Γιατί σίγουρα πρόκειται για πολλά τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξετάζουν όλες αυτές τις διατάξεις της ε, γλωσσικής νομοθεσίας της Σλοβακίας. Τώρα τόσο εσείς όσο και ε, εμείς από την Επιτροπή πολλές φορές έχουμε συναντηθεί με διάφορους εκπροσώπους τόσο από τη Σλοβακία όσο και από την Ουγγαρία. Έχουμε... Έχουν φτάσει σε εμά χιλιάδες μηνύματα για αυτό το θέμα από ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο από τις δύο αυτές χώρες, Σλοβακία και Ουγγαρία δηλαδή. Στις συζητήσεις που είχαμε με εκπροσώπους και από τις δύο αυτές χώρες, ξεκαθαρίσαμε από τη δικιά μας την πλευρά ότι η εφαρμογή των διατάξεων, πέρα από την ανάλυση που θα κάνει η Επιτροπή, η εφαρμογή του νόμου αυτού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η εφαρμογή αυτή, η θέση σε ισχύ δηλαδή, πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία. Στηρίξαμε επίσης, είπαμε δηλαδή ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε ε, τη Σλοβακία ώστε να βρεθούν οι λύσεις που πρέπει. Η κοινή δήλωση εξάλλου που υπέγραψαν οι δύο πρωθυπουργοί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος και αποτελεί και εγγύηση πιστεύω για το ότι τελικά θα βρεθεί μια αποδεκτή και από τις δύο πλευρές λύση. Για την κυρία Τρούπελ τώρα. Η συνεργασία μας με χώρες που μοιάζουν όσον αφορά την ε, γλωσσική ποικιλομορφία είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αναφερθήκατε στην Κίνα, δεν είναι μόνο εκεί, είναι και αλλού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε παρόμοιες καταστάσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, ώστε να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλο και περισσότερα πανεπιστήμια στα διάφορα κράτη-μέλη, πανεπιστήμια λοιπόν που προωθούν την εκμάθηση γλωσσών όπως είναι τα Ινδού, τα γλώσσα των Μανταρίνων, Κινέζικα, είναι ευκαιρίες αυτές που προσφέρονται στους φοιτητές των πανεπιστημίων αυτών. Και εμείς έχουμε ανταποκριθεί θετικά στις πρωτοβουλίες αυτές. Δεν θα περιοριστούμε όμως μόνο σε αυτή την πτυχή αμοιβαία πρόθεσης, δηλαδή της εκμάθησης ξενογλωσσών, γιατί κάθε φορά που έχουμε διάλογο, θέλουμε πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε την άλλη πλευρά, αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε να προωθήσουμε τις δικές μας αξίες, δηλαδή ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια βασική αξία για μας. Ποτέ δεν ξεχνάμε να αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα. Ποτέ δεν το παραλείπουμε. Ακόμα κι αν κάποτε αποδεικνύεται πολύ δύσκολο. Παρ' αυτά, κάθε φορά που έχουμε διάλογο με τους εταίρους μας, είτε στην Κίνα είτε αλλού, το βάζουμε αυτό το θέμα. Και μας απαντάνε πάντα, ναι, το έχουμε στην ημερήσια διάταξη, ναι. Ακόμα και όταν πρόκειται για την πολυγλωσία, να ξέρετε ότι αποτελεί μέρος του, της πρόθεσης του πολιτισμικού διαλόγου. Στον κύριο Τάκουλα Πρώτα απ' όλα, κύριε Τάκουλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την θετική αξιολόγηση που κάνατε του έργου μου. Και χαίρομαι επίσης για το ότι κάποιος που γνωρίζει τόσο καλά τα πράγματα, με βαθμολογεί τόσο καλά. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος Μπαρόσο ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας εντολής θα υπάρχει υπεύθυνο επίτροπος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Θα είναι ένα επίτροπος ο οποίος θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Ελπίζουμε σύντομα να έχει επικυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και να αρχίσει να ισχύει, Οπότε το χαρτοφυλάκιο αυτό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μάλλον ε, η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων θα αρχίσει να ισχύει συγχρόνως. Αυτή θα είναι μια νέα εξέλιξη. Θα ενισχύσει τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οι αρμοδιότητές μας θα είναι περιορισμένες και στο μέλλον. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Το θέμα αυτό θα αναλύεται όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, όπως σας έλεγα και πριν, και στα πλαίσια ε, του διαλόγου που έχουμε με τρίτες χώρες, είτε είναι ευρωπαϊκές είτε δεν είναι. Στην κυρία Νεμπεμπάλοβα τώρα. Η πρόθεση της γνώσης της γλώσσας των μεταναστών είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, χώρες μέλη όπου οι αρχές επιμένουν να προωθήσουν την μητρική γλώσσα των μεταναστών. Βέβαια ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες γλώσσες μεταναστών στην ε, Ευρώπη. Όμως, Πρώτα απ' όλα πρέπει να μαθαίνουν οι μετανάστες την γλώσσα της χώρας υποδοχής. Είναι λεπτό το ζήτημα βλέπετε γιατί σε μερικές χώρες, σε μερικές πρωτεύουσες, τι μας είπαν. Καλύτερα μην το θίγετε αυτό το ζήτημα γιατί είναι ένα θέμα καυτό. Πάρα πολύ λεπτό πολιτικά. Αλλά ακόμα και έτσι, η θέση μας είναι σαφής. Εμείς πιστεύουμε ότι πέρα από την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, που σίγουρα αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την ε, ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να σεβόμαστε και τις μητρικές γλώσσες των μεταναστών. Οι ειδικοί λένε ότι αν δεν γνωρίζεις καλά τη μητρική σου γλώσσα, δεν μπορείς να μάθεις καμία άλλη γλώσσα καλά. Και αυτό, για να μην επαναλάβω αυτό που έλεγα και πριν, για τον ρεαλισμό που πρέπει να διέπει την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Τα διάφορα μοντέλα ένταξης που γνωρίζουμε διαφέρουν μεταξύ τους κατά πολύ. Έχουμε ολόκληρο κατάλογο με βέλτιστες πρακτικές από διάφορες χώρες μέλη. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία, αλλά και άλλες χώρες που έχουν τέτοια παραδείγματα συστημάτων ένταξης αυτά, αυτές οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να διαδίδονται και να εφαρμόζονται και αλλού. Όσον αφορά τώρα την εκμάθηση ξένων γλωσσών όσο πιο νωρί γίνεται, όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά, πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγινα από το ενδιαφέρον που έχει ξεσηκώσει η πρωτοβουλία μας αυτή. Υπάρχουν ερευνητές, ειδικοί, καθηγητές πανεπιστημίων πάρα πολύ γνωστοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν στηρίξει την πρωτοβουλία μας αυτή και θα συμμετάσχουν. Βέβαια, τα κράτη-μέλη πρέπει και τα ίδια να βοηθήσουν. Ο πολιτικός διάλογος, πιστεύω, θα βοηθήσει ώστε να συμμετάσχουν και τα κράτη-μέλη στην πρωτοβουλία αυτή. Συνεχίζω για τα ουαλικά, Ιρλανδικά. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι το εξής. Είχα επαφές με τις Ιρλανδικές αρχές και μπορώ να σας πω ότι οι Ιρλανδικές αρχές αναλύουν τη δικιά μας δουλειά. Την παρακολουθούν στενά υπήρξε μια έκθεση που δεν μπορέσαμε έγκαιρα να την μεταφράσουμε στα Ιρλανδικά και η αντίδραση των Ιρλανδικών αρχών ήρθε αμέσως. Σήμερα λοιπόν η συμπερίληψη της γλώσσας αυτής στα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα έχει προχωρήσει πολύ. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν φτάνει να κάνουμε εμείς προσπάθειες, στα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα, αν από την άλλη μεριά η Ιρλανδία δεν έχει αρκετούς γλωσσομαθείς, δεν έχει αρκετούς νέους που να ξέρουν ξένες γλώσσες. Γιατί πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση, πώς θα ανταποκριθούμε στη ζήτηση που έχουμε και όσον αφορά τη διερμηνία και όσον αφορά την μετάφραση εγγράφων ή τα επίσημα έγγραφα τα οποία πρέπει να μεταφράζονται και στα Ιρλανδικά καταλαβαίνετε ότι είναι μια δουλειά που δεν γίνεται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα απ' όλα γίνεται από το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με την Ιρλανδική γλώσσα. Βλέπετε, όλος παραδόξος έχει να κάνει με γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ και στα κοινοτικά όργανα. Τα αγγλικά, τα γαλλικά, πρόσφατα ξεκινήσαμε προγράμματα ώστε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία να πείσουμε τους νέους ότι πρέπει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Αλλιώς, για να είμαστε ειλικρινείς, αν ε, δεν γίνει αυτό, τα ευρωπαϊκά κοινωτικά όργανα δύσκολο θα μπορέσουν να καλύψουν τις γλώσσες στο μέλλον. Τα επόμενα 5-10 χρόνια δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα με τις μεταφράσεις. Για τα αγγλικά είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και θα σας δώσω παράδειγμα. Για τα γαλλικά ο αριθμός διερμηνέων που θα έχουμε τα επόμενα 10 χρόνια θα μειωθεί στο ίμιση. Αν δεν φροντίσουν οι γαλλικές αρχές να κάνουν από την πλευρά τους προσπάθειες για να αυξήσουν τον αριθμό αυτό. Διότι, σας είπα, δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε διερμηνία σε όλες τις συνεδριάσεις που χρειάζονται. Θα έχουμε διερμηνία μόνο σε περιορισμένες συνεδριάσεις. Αυτό είναι ο κίνδυνος και αυτές είναι και οι προκλήσεις που έχουμε για το μέλλον. Άρα δεν ισχύει μόνο για τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες, Όσο και αφορά τώρα την πρωτοβουλία του Προέδρου Μπαρόσο για την ε, νεότητα σε κίνηση, Youth in Move, είναι μια πρωτοβουλία πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, ξεκινάει, πρέπει δηλαδή να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και να έχουμε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει της πρότασης της Επιτροπής, για να δούμε τι λένε και αυτοί. Τέλος, να απαντήσω στην κυρία Παλιαδέλη. Αναφέρθηκα λίγο πριν στο ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με την τέος Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όλο και πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι η λύση για το θέμα του ονόματος και την ε, γλώσσα της χώρας, είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την χώρα αυτή όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής της. Η τελευταία ερώτηση, και ίσως να είναι και πιο δύσκολη από όλες, ήταν πώς ξέρουμε κατά πόσο πρόκειται για μια γλώσσα ή για μια διάλεκτο. για αυτό το θέμα μπορώ να σας πω ότι αυτό τελικά είναι θέμα επικουρικότητας. Είναι δηλαδή μία απόφαση που την παίρνουν οι αρχές των χωρών μελών και των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δικιά τους αποκλειστική αρμοδιότητα. Πολλές φορές εγώ ρώτησα τους ειδικού για να ξέρω, για να μπορώ να κάνω τη διάκριση της διαλέκτου από μία γλώσσα. Και μου είπαν ότι τελικά τη διαφορά την κάνουν οι πολιτικοί και όχι οι δικοί και οι πυρογνώμονες. Θα σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το θέμα της γλωσσικής πολυμορφίας είναι παλιό θέμα και σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Διαπιστώνω και εγώ ότι θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε αρκετούς διερμηνείς. Προωθούμε την ιδέα της γλωσσικής πολυμορφίας. Έχουμε δεσμευτεί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε μια έλλειψη διερμηνέων. Γιατί βεβαίως υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία που δεν μπορεί πλέον να τροφοδοτήσει την αγορά με όσους διερμηνείς και μεταφραστές χρειάζονται. Βλέπετε λοιπόν ότι αν θέλουμε όντως να υπάρχει πολυγλωσία στην Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρχουν και άτομα τα οποία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα αυτό. Θα πρέπει ίσως τα εθνικά κοινοβούλια να συζητηθεί αυτό. Εμείς στην Γερμανία, στον Bundestag, λέμε διαρκώς ότι πρέπει να στηρίξουμε την γερμανική γλώσσα. Και δεν αναρωτιόμαστε πάντα αν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν την μετάφραση και την διερμηνία της γερμανικής γλώσσας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας κύριε Επίτροπε και πραγματικά ξέρουμε ότι εμείς στα εθνικά μας κοινοβούλια πρέπει να κάνουμε δουλειά. Και βεβαίως οι αγγλόφωνοι, καθότι η αγγλική γλώσσα είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη γλώσσα στην Ευρώπη, δεν έχουν ίσως τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εγώ όμως που ε, είμαι Γερμανίδα και έχω λάβει εντολές συγκεκριμένες από τον πρόεδρο του Bundestag, θέλω να στηρίξω τη δική μου γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ελπίζω ότι θα ξανάρθετε. Τα τελευταία τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια ήσασταν σε αυτή τη θέση. Σας ευχαριστούμε γιατί σε πολλούς τομείς κινήσατε τα πράγματα, δεσμευθήκατε και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε και μας μιλήσατε στην Επιτροπή Πολιτισμού. So, liebe Kolleginnen und... Συνάδελφοι, μην κουνηθείτε από τις θέσεις σας, σας παρακαλώ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα. Πρόκειται για την παρουσίαση των βραβείων. Σας το διαβάζω σε αγγλικά. Πρόκειται για το βραβείο το ευρωπαϊκό του Κάρλο Μάγλου, το οποίο ξεκίνησε το 2008 σαν μια κοινή πρωτοβουλία του βραβείου Σαγλωμάν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει μακριά παράδοση. Με τον πρόεδρο Πέτερινγκ λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Σκοπός αυτού του βραβείου είναι να βραβεύσει σχέδια νέων 16 με 30 ετών είναι αυτοί οι νέοι και να προωθήσουν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατανόηση. Και βεβαίως πρόκειται για σχέδια τα οποία υποβάλλονται από κοινού από νέους που προέρχονται από πάνω από μία χώρα μέλη. 200 τέτοια προγράμματα και σχέδια υποβλήθησαν το 2009 και Βεβαίως υπήρχαν δύο ε, στάδια επιλογής και αξιολόγησης. Πρώτον σε μια εθνική επιτροπή, όπου υπήρχαν και δύο ευρωβουλευτές και ένας εκπρόσωπος μιας οργάνωσης χρηστών. Το δεύτερο επίπεδο αξιολόγησης και επιλογής είναι μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μέλη με Ευρωπαίους βουλευτές, ευρωβουλευτές και μέλη του Ιδρύματος Σαγλεμάνια. Ο Καρλ Σμιτ ήταν μέλος αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Άχεν στις 19 Μαΐου έλαβε χώρα η τελετή απονομής. Η τρίτη επιλογή, το τρίτο βραβείο, είναι ένα γερμανικό σχέδιο το οποίο λέγεται Oberkante Unterlippe Και δεν ξέρω αν αυτό μεταφράζεται. Oberkante Unterlippe. Πρέπει να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα project, ένα πρόγραμμα το οποίο υπευλήθη από νέους μια ένωση, ένα σύλλογο νέων, οι οποίοι είναι Γερμανοί. Το δεύτερο βραβείο δόθηκε σε μια γαλλική θεατρική ομάδα από την πόλη του Αλμπί. Πρόκειται για μια σχολή που βρίσκεται στο Αλμπί, θεατρική, και το πρώτο βραβείο 5.000 ευρώ. Το πήρε η Πολωνία, ένα σχέδιο από την Πολωνία, Europe Needs You είναι ο τίτλος. Το υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Φόρουμ IG. Και βεβαίως έχουμε εδώ τρεις νέους από αυτήν την ομάδα, την κυρία Λάρα Σέπελ, που εκπροσωπεί τη Γερμανία. Κάπου είναι, πίσω, στα έδρανα. Την κυρία, την Δεσποινίδα Μαρή Τεριέ, που εκπροσωπεί τη Γαλλία, και την Χίλτε Ντελόε, που εκπροσωπεί την Πολωνία. Είναι η κυρία που βρίσκεται δίπλα μου. Και επειδή κέρδισαν το πρώτο βραβείο, θα τους δώσουμε και λίγα λεπτά να μας παρουσιάσουν το διαγωνισμό. Okay, dear all, I'm really, really grateful Σας ευχαριστώ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιον σας. Είναι, είμαι αρκετά αγωμένη πρέπει να σας πω και θα ήθελα σε 10 λεπτά να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμά μας, το Europe Needs You, ε, που κέρδισε το βραβείο του Καρλομάγνου για το 2009 και πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι που δείχνουν την πιστοσύνη στο πρόγραμμα αυτό. Χάρη στο βραβείο συνεχίζουμε με ένα δεύτερο κύκλο για το επόμενο, τον επόμενο χρόνο. Υπάρχει το πρόγραμμα από τον Ιανουάριο του 2008 και αναπτύχθηκε το πρόγραμμα το πρώτο ήμιση του έτους, ε, συνέχισε να λειτουργεί ένα έτος και περνάμε σε έναν επόμενο χρόνο. Ονομάζομαι Χίλντε Τελέου, είμαι από τις κάτω χώρες Ε, περιλαμβάνονται φοιτητές ε, στο πρόγραμμα μας από 43 χώρες ολόκληρη την... Ε, δηλαδή από όλη την Ευρώπη είναι φοιτητές από διάφορες εθνικότητες. Εμείς ήρθαμε, στην αρχή ξεκινήσαμε με έξι άτομα. Έξι μόνο άνθρωποι ήμασταν στην αρχή. Εδώ υπάρχουν και εικόνες ανθρώπων που ήδη είχαν ε, συμμετάσχει και τώρα και αυτή τη στιγμή έχουμε 240. Αρχικά λοιπόν προήλθαν από την Ισπανία, ε, συναντηθήκαμε έτσι ώστε στα γυμνάσια μας μάλλον με την ιδέα ότι στα γυμνάσια μας δεν είχαμε αρκετά ευρωπαϊκά θέματα στην εκπαίδευσή μας και θεωρήσαμε πως η νέα γενεά που θα αποτελέσει τους μελλοντικού ηγέτες και τους ανθρώπους που θα πιάσουν τα ψηλά πόσα στην Ευρώπη, γι' αυτό και θα έπρεπε να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για τα ευρωπαϊκά θέματα. Και θελήσαμε να τους δώσουμε μια ευκαιρία να δουν τι ιδέες υπάρχουν ήδη, δηλαδή να μπορέσουν ε, οι μαθητές των ε, σχολείων στην Ευρώπη, των γυμνασίων, να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρώπη. Γι' αυτό κάναμε μια έρευνα πρώτα στην Ευρώπη, δηλαδή πώς γίνεται η εκπαίδευση. Ήταν μια έρευνα που έγινε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά, ότι δηλαδή Όλα είναι και περισσότεροι μαθητές αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα και το έβλεπαν, ότι δηλαδή η εκπαίδευση δεν ασχολείται με τα θέματα που απασχολούν τις Βρυξέλλες δεν γνώριζαν καν τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τον κόσμο και ιδιαίτερα για τους νέους. Η σχετική εκπαίδευση λοιπόν ήταν πολύ επιφανειακή και υπήρχε και μια στάση απέναντι στην Ευρώπη ότι δηλαδή είναι πολύ μακριά από μας, είναι κάτι το κατανόητο για μας, ήταν γενικά διάφοροι για την Ευρώπη. Αυτό επίσης σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν είναι πραγματικά δραστήριοι στην ε, κοινωνία. Δεν ασχολούνται με τίποτα εθελοντικά προγράμματα, για παράδειγμα, οι ανταλλαγέ και υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Υπάρχουν ε, διάφορα προγράμματα, όπως αυτό που μόλις είπατε για το Youth on the Move, ε, όμως γίνει γεγονός ότι τα, οι, οι νέοι δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις δυνατότητες. Και επειδή δεν γνωρίζουν και αδιαφορούν και αδιαφορούν επειδή δεν γνωρίζουν, ε, και καθώς οι νέοι αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης, θέσαμε αυτό το στόχο, να δώσουμε δηλαδή περισσότερες δυνατότητες στους μαθητές ολόκληρη την Ευρώπη. Θέσαμε το στόχο ότι να βελτιώσουμε τις πρακτικές γνώσεις για την Ευρώπη, ώστε να υπάρχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του προγράμματός μας και να αυξήσουμε την, αλλαγή, την ανταλλαγή πληροφοριών για τις δυνατότητες για τους ε, μαθητές των γυμνασίων. Και αυτό μέσω σεμιναρίων, όπου πηγαίναμε στα, και εργαστηρίων. Πηγαίναμε δηλαδή στα διάφορα σχολεία, του είπαμε τα όσα ξέρουμε, πώς ταξιδεύουμε, τι είδους δυνατότητες ανταλλαγών υπάρχουν, αλλά και επίση μια εισαγωγή για την ιστορία ιστορία της Ευρώπης, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Με αυτές λοιπόν τις πληροφορίες και αυτές τις πρακτικές γνώσεις που είχαν οι μαθητές ε, μπόρεσαν να οργανώσουν κάποιες δράσεις για τα σχολεία τους και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για ένα εργαστήριο και ένα σύντομο βίντεο που θα σας δείξω να, δηλαδή θέλαμε να δώσουμε κίνητρα στους νέους ώστε να ενημερώσουμε τη σειρά τους και άλλους φοιτητές, άλλους μαθητές. Όλοι είμαστε εθελοντές, δηλαδή και εμείς ζητάμε τους άλλους, από τους άλλους μαθητές να πάνε σε άλλο σχολείο και να πούν ε, τι έμαθαν. Στην αρχή είχαμε πρόβλημα με τα σπόρους και αλλά μετά είπαμε εντάξει δεν μας νοιάζει και πολύ. Αυτό που θέλαμε να προωθήσουμε ήταν να ε, σπρώξουμε τους μαθητές, ε, να, να τους κινητοποιήσουμε. Πολλά εργαστήρια, διαλέξεις σε ένα σορμέρι και επίσης κάναμε και εργαστήρια εκπαίδευσης, κατάρτισης, όπου τους μάθαμε να πηγαίνουν στα σχολεία και να κάνουν και εκείνοι με τη σειρά τους ε, άλλα παρόμοια εργαστήρια με παιχνίδια, συζητήσεις. εδώ μια από τις εικόνες ε, μιας ε, από τις ε, ενός από τα εργαστήρια κατάρτισης. Επίσης συγκεντρώσαμε ένα σωρό ιδέες για παιχνίδια, συζητήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία και άρα τα παιδιά πήγαιναν στα σχολεία τους, στα διάφορα γυμνάσια και πήγαιναν σε δύο-τρεις τάξεις για να διαδώσουν ε, τις ιδέες. Και μέσα από αυτό το χάρτη βλέπετε τώρα πόσο έχει απλωθεί το πρόγραμμά μας. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που ήθελα να σας δείξω. Δεν θέλει όμως να εμφανιστεί. Okay. Is there no music? Okay. Well, at least you have an idea like how students were. Um, Τουλάχιστον βλέπετε, έχετε μια εικόνα για το πώς συνεργάζονταν ε, τα παιδιά. 15 ετών είναι οι μαθητές αυτοί, είναι στις κάτω χώρες. Έχω πάει και σε ένα σχολείο στην Πολωνία μαζί με Πολωνούς ε, μαθητές. Of that aspect of Οπότε υπάρχει και αυτή η πτυχή της πολυγλωσσίας. Project in, in Polish and English or in Spain and English or in German and English. And um, the action they did for their school was... Um, Και η δράση που κάναμε στο δικό του σχολείο ήταν να ζωγραφίσουν διάφορα στερεότυπα που έχουν στο μυαλό τους για κάθε χώρα της Ευρώπης. Okay. No, It's okay. Ah. Okay, this is such a pity, but I uh, hope you had a really short idea how it was looking like. Μια σύντομη ιδέα λοιπόν, μια σύντομη εικόνα για το τι γίνεται. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Τα παιδιά είχαν μεγάλη διάθεση, θέλαν να φτιάξουν μια ζωγραφιά. με με τον ενθουσιασμό των παιδιών έδειξαν στο σχολείο ότι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη. Και ακολούθησαν μετά αυτή την ιδέα με τη βοήθεια των ε, δασκάλων τους. Δεκαεννιά χώρες, 200 ε, παιδιά έχουν καταρτιστεί και μέσω των εργαστηρίων φτάνουμε σε πολλούς νέους, αλλά δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε, γιατί κάποιες φορές είναι μια τάξη 20 παιδιών, ενώ άλλες φορές είναι μια παρουσίαση για ένα ολόκληρο σχολείο. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό, αλλά η ιδέα είναι πάντοτε η ίδια. Να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Και έχουμε και άλλες ιδέες. Αυτή τη στιγμή, φέτος, δουλεύουμε φτιάχνοντας επιστολές ώστε να έρθει κόσμος να τους καλέσουμε στο... να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες, ακόμα και βουλευτές, ευρωβουλευτές θέλουμε να συναντήσουμε, έχουμε φτιάξει και ένα δίκτυο, εδώ βλέπετε το δίκτυό μας. και έτσι μπορούν να συνδεθούν και οι μαθητές από τις διάφορες χώρες, μπορούν εύκολα να βρουν η μεν δε. Και πάλι λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω που δείξατε εμπιστοσύνη σε αυτό το πρόγραμμα στο ε, Europe Meet You. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνδεθούμε και απόψε υπάρχει ένα πραγματικά ωραίο πρόγραμμα για τους ε, νικητές του βραβείου και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Hilde. Ευχαριστώ πολύ την Χίλντε. Είναι ένα ωραίο συμπλήρωμα του Κοινοβουλίου των Νέων. Έχουμε δύο τέτοια κοινοβουλία, σας το επιθυμίζω αν δεν το ξέρετε, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς όχι, εσείς το κάνατε μόνοι σας, ήταν δική σας πρωτοβουλία και αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για το Κομίνιος, για τα βραβεία που δίνονται και εκεί. Ίσως λοιπόν μπορείτε και εκεί να έρθετε σε επαφή και να χρηματοδοτηθείτε κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε μήπως αυτό είναι δυνατό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι δημιουργήσατε μια ωραία κοινότητα, ένα δίκτυο το οποίο θα πολλαπλασιαστεί. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Μαρή Τεριέ. καλημέρα σας. Θα σας μιλήσω γαλλικά, αλλά η παρουσίασή μου είναι στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μας προσκαλέσατε εδώ και είμαι πολύ περήφανη που μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω το φεστιβάλ Ακτέα. Φεστιβάλ που κάνει εκδηλώσεις στο δρόμο και προσφέρει παραστάσεις θεατρικές. Εγώ είμαι η Μαρή Τεριέ, είμαι υπεύθυνη για θέματα επικοινωνίας του φεστιβάλ αυτού. Το φεστιβάλ Ακτέα ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια με περίπου 10 άτομα. Σήμερα είμαστε 30 φοιτητές της Σχολής Μηχανικών της πόλης του Αλμπή και πραγματικά είμαστε όλοι εθελοντές και χρησιμοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας για να οργανώσουμε αυτό το φεστιβάλ. Κάθε χρόνο καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έρχονται στην πόλη του Αλμπή και μοιράζονται μαζί μας το πάθος μας για το θέατρο και την Ευρώπη. Τι είναι το Άκτεα λοιπόν. Είναι ένα φεστιβάλ θεατρικό το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Είναι το θεατρικό φεστιβάλ με θειάσους φοιτητικού από όλη την Ευρώπη. Καταρχήν ανεβάζουμε ένα γαλλικό έργο και ένα ξένο έργο. Ο καθένας βέβαια, ε, ο κάθε ηθοποιός παίζει στη μητρική του γλώσσα. Έχουμε δύο επιτροπές, μία που αποτελείται από επαγγελματίες και μία από ερασιτέχνες. Στο τέλος, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, έχουμε μία τελευταία παράσταση και παράλληλα με το επίσημο, αν θέλετε, φεστιβάλ θεάτρου, έχουμε το φεστιβάλ OFF, το ανεπίσημο, το οποίο, αν θέλετε, κάνει παραστάσεις και εκδηλώσεις στο δρόμο. Το Ακθέα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ στην μικρή πόλη του Αλμπί. 60.000 κατοίκους μόνο έχει στην Νότια Γαλλία η πόλη του Αλμπί. Και έχει μία σχολή μηχανικών, ένα πανεπιστήμιο, αλλά πολλά μικρά παιδιά. Είναι λοιπόν σημαντικό για την πολιτιστική ζωή της ε, πόλης και της περιοχής και την ενημέρωση για την Ευρώπη. Είμαστε πολύ περήφανοι λοιπόν που κερδίσαμε αυτό το δεύτερο βραβείο, το οποίο μας στηρίζει, μας ενθαρρύνει και την ίδια ώρα πήραμε και το μετάλλιο, το δημοτικό μετάλλιο της πόλης του Αλμπή. Αυτό είναι για μας μια επιπλέον αναγνώριση. Κάθε χρόνο λοιπόν, στις διακοπές του Πάσχα, το φεστιβάλ λαμβάνει χώρο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Τα παιδιά λοιπόν είναι σε διακοπές. Μπορούν λοιπόν ακόμα και άτομα τα οποία δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν στο θέατρο να έρθουν και να δουν τις παραστάσεις. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο η ομάδα που οργανώνει το φεστιβάλ συναντιέται πολύ περισσότερο το Μάρτιο και τον Απρίλιο βέβαια γιατί πρέπει να στηρίξουμε την οργάνωση του φεστιβάλ, καλούμε καλλιτέχνες, φοιτητές από όλη την Ευρώπη και αυτό βεβαίως χρειάζεται οργάνωση. Πρέπει να έρθουν, πρέπει να τους βρούμε δωμάτια, να οργανώσουμε το που θα φάνε, δεν μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το τηλέφωνο και το mail για να οργανώσουμε όλες αυτές τις επισκέψεις. Το θέατρο είναι ένα αληθινό θέατρο και η είσοδος είναι ένα ευρώ. Είναι ένα συμβολικό εισιτήριο γιατί πραγματικά θέλουμε να προσελκύσουμε πολύ κόσμο. Ιδίως νέους από δύσκολες περιοχές στα περίχωρα της πόλης του Αλμπή, άτομα που συνήθως δεν έχουν μεγάλη σχέση με το θέατρο και τους ζητάμε κατόπιν να παραμείνουν μετά την παράσταση γιατί οι καλλιτέχνες οργανώνουν συζητήσεις με το κοινό, με τους φοιτητέ και με όλους τους θέατες έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική ανταλλαγή ε, και συζήτηση. Το παράλληλο φεστιβάλ, το φεστιβάλ OFF, το ανεπίσημο, λαμβάνει χώρα στην πόλη του Αλμπί, ως ένα βαθμό και στο Πανεπιστήμιο, γιατί θέλουμε να είμαστε σε στενή επαφή και με τους άλλους φοιτητές, και σε μια πλατεία της πόλης του Αλμπί, στην πλατεία Σαν Σεσίλ, που είναι μια κεντρική πλατεία. Θέλουμε πραγματικά να έρθουμε σε επαφή με άτομα που συνήθως δεν πάνε στο θέατρο και δεν βλέπουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Έχουμε και μία μέρα που αφιερώνεται στα παιδιά, πλησιάζουμε δασκάλους, βρεφικούς, ε, παιδικούς σταθμούς και με μεγάλη χαρά κάθε χρόνο βλέπουμε παιδιά τα οποία ακόμα και δεν καταλαβαίνουν πάντα τη γλώσσα της παράστασης, ε, βλέπουν τους καλλιτέχνες, τους κλόν, τους ακροβάτες και συμμετέχουν με το γέλιο τους σε αυτό το φεστιβάλ. Πρόκειται για μας, για μια ολόκληρη εβδομάδα πολιτιστική. Στη σχολή μας προσκαλούμε και φιλοξενούμε περίπου 100 ε, καλλιτέχνες κάθε χρόνο. Έχουμε καλλιτέχνες από όλες τις χώρες. Και πολλές φορές βλέπουμε καλλιτέχνες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο φεστιβάλ να ξαναέρχονται ακόμα και αν δεν συμμετέχουν, για να είναι παρόντες την εβδομάδα του θεατρικού φεστιβάλ. Επαναλαμβάνω ότι ο κάθε θείασος χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, κάτι το οποίο τους υποχρεώνει για να γίνουν κατανοητοί από ένα κοινό που πολλές φορές δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα, να χρησιμοποιούν γλώσσα του σώματος, κινήσεις, χειρονομίες, οι οποίες τους κάνουν πιο κατανοητούς με πολύ συμβολική σκηνοθεσία. Το βραβείο Καρλομάγνου είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών και της δουλειάς μας. Πέρσι αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες για την οργάνωση του φεστιβάλ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ζούμε χάρη σε επιδοτήσεις, και πολλές επιχειρήσεις μείωσαν τη στήριξη. Ε, πολλές φορές λοιπόν ε, έχουμε δυσκολίες να προσελκύσουμε ξένους θειάσους γιατί τους φιλοξενούμε, τους προσφέρουμε φαγητό και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι θείασοι δεν μπορούν να έρθουν χωρίς αυτή την οικονομική στήριξη. Βεβαίως κάνουμε διαφήμιση και φέτος για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι φοιτητέ που είχαν ακούσει ότι πήραμε το βραβείο Σαλομάνι μας ζήτησαν να έρθουν και να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ για φέτος. Επίσης αποφασίσαμε ότι ένα τμήμα των παραστάσεων θα πρέπει να μεταφραστούν, γιατί τα μικρά παιδιά κυρίως πολλές φορές έχουν δυσκολία να παρακολουθήσουν ε, τις παραστάσεις. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν καλύτερα ε, το σενάριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, Marie. Vous avez Ευχαριστώ πολύ τη Μαρή. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ δημιουργικό πρόγραμμα. Ελπίζω να συνεχίσετε εσείς οι επόμενοι, γιατί εσείς κάποια στιγμή θα τελειώσετε τις σπουδές σας. Αλλά αν πρόκειται για τέτοια σχολή ε, μηχανικών Η κυρία Σόπε έχει το λόγο για το τρίτο βραβείο. Γεια σας, το όνομά μου είναι Λάρα Σόπε, είμαι από τη Γερμανία και είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι Ε, μεγάλη ευχαρίστηση. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να κάνω την παρουσίασή μου στα γερμανικά. Ist der Name der ganzen, des ganzen Projektes. Und dies ist ein mehrdeutiger Titel für ein ökologisches Unternehmen. Πρόκειται για μια οικολογική προσπάθεια Απευθυνόμαστε σε μαθητές, φοιτητές από την Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία και Ολλανδία. Και πρόκειται για ένα πρόγραμμα μιας πιο σφαιρικής πολιτικής διάστασης. Το όνομα Oberkante Unterlippe ουσιαστικά σημαίνει ότι το ποτήρι είναι γεμάτο, ότι φτάνει πια και ουσιαστικά αναφέρεται σε ύδατα τα οποία φτάνουν σε κάποιες λεκάνες, σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, δημιουργώντας πλημμύρες και βεβαίως εδώ αναφερόμαστε και στη βιομηχανική μόλυνση. Το Oberkante Unterlippe χαρακτηρίζει επίσης και μια μελέτη περιφερειακή στην περιοχή αυτή του παραπόταμου του Ρήνου, γιατί Λίπε είναι ένας παραπόταμος του Ρήνου. στην Ρενανία Βεσφαλία, είναι περιοχή αυτή, και είναι πολύ συγκεκριμένη η εμπλοκή των ε, τοπικών αρχών, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών αρχών. Το Σεπτέμβριο του 2007, 12 μαθητές ξεκίνησαν αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για μαθητές ενός γυμνασίου γερμανικού συνεργασία που οδήγησε μαθητές από την Ολλανδία και την Πολωνία να συνεργαστούν μαζί τους. Το ερώτημα ήταν υπάρχουν τοπικές απαντήσεις σε παγκόσμια προβλήματα και εδώ ήταν ένα καθαρό οικολογικό πρόβλημα και αποδείξαμε ότι βεβαίως η παγκοσμιοποίηση έχει συνέπειες τοπικές που αφορούν και πλήττουν άτομα συγκεκριμένα. Αλλά και ότι υπάρχει και μία δυνατότητα δράσης ατομική, συλλογική, σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε τις προσπάθειές μας λέγοντας ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και φταίει η παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε να δεσμευτούμε σε τοπικό επίπεδο για να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Όσον αφορά λοιπόν τον κίνδυνο της πλημμύρας, είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, γι' αυτό και δημιουργήσαμε εταιρικέ σχέσεις μεταξύ σχολείων και γυμνασίων της περιοχής. Η εικόνα που βλέπετε στην οθόνη είναι και βασίζεται σε μια βασική ιδέα ότι σε ένα τμήμα της γης υπάρχει λειψιδρία και σε άλλα μέρη της γης υπάρχουν πλημμύρες. Υπάρχει πολύ νερό. Βλέπετε αυτές τις εικόνες, είναι εικόνες του ποταμού Λίπε. Αυτό είναι το ποτάμι που μας απασχόλησε. Είναι ένα ποτάμι, όπως σας είπα και προηγουμένως, παραπόταμος του Ρήνου. Βλέπετε τις εικόνες. Εδώ βλέπετε διάφορα έργα που γίνονται στις όχθες του ποταμού Λίπε για να αποφευχθεί η υπερχείληση. Και βεβαίως εδώ έγιναν διάφορα έργα στις δύο όχθες και η δημιουργία καναλιών. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι το νερό, το επίπεδο του νερού ανεβαίνει, αυξάνεται. Προσπαθήσαμε να διοχετεύσουμε αυτό το νερό αριστερά-δεξιά με τη δημιουργία ε, κάποιων καναλιών. Εδώ δηλαδή οι δυνατότητες αυτές δεν υπήρχαν και δημιουργήθηκαν. Το νερό κυλάει πλέον σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και δεν χάνεται. Και εδώ βλέπετε τις συγκεκριμένες προσπάθειες που κάναμε. Οδηγήσαμε αν θέλετε, καταρχήν τους ειδικού στην ειδική προσοχή που πρέπει να δοθεί στην πανίδα, τη χλωρίδα. Πολλές κατηγορίες ψαριών, παραδείγματος χάριν, που κινδύναβαν να εξαφανιστούν. Είδαμε παραδείγματος χάρη ότι πολλά είδη που είχαν εξαφανιστεί επανήλθαν μετά τα έργα που έγιναν. Και αυτό είναι δείγμα ότι το ίδιο και αυτά τα έντομα τα οποία βλέπετε εδώ πρόκειται για έντομα παραδείγματο χάρη που έρχονται από την Αφρική και την Νότια Ευρώπη τα οποία υπήρχαν και στην Νότια Γερμανία Σήμερα τα βρίσκουμε και στην περιοχή μας. Αυτό είναι βεβαίως δείγμα ότι υπάρχει και υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι νέα είδη. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι εργαστήκαμε όλοι μαζί οργανώνοντας ένα συνέδριο με τη συμμετοχή βεβαίως και των γονέων, πολιτικών και άλλων προσωπικότητων. με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αναρωτηθήκαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τι σχέση έχουμε με την Ευρώπη, πώς βλέπουμε το μέλλον μας σαν Ευρωπαίοι, τι άγχη μας δημιουργεί η Ευρώπη, η αλλαγή του κλίματος. Και από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το συμπόσιο, σε αυτό το συνέδριο, διατυπώσαμε κάποιες προτάσεις και κάποιες ιδέες όσον αφορά την παρόμοια, αν θέλετε, αντιμετώπιση ε, φαινομένων πλημμύρας, και υπερχείλησης των υδάτων και σε άλλα ποτάμια και σε άλλες περιοχές. Αυτά. Εδώ βλέπετε όλους ε, τους ε, μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τη Λάρα, λέει η Πρόεδρος. Πολύ καλή ιδέα είχατε. Νέα παιδιά τα οποία εδώ προσπαθούν να βρουν λύσεις για τα σφάλματα και τις καταχρήσεις και την υπερεκμετάλλευση των γονιών τους, των παππούδων τους και των προπαππούδων τους. Έχετε δίκιο ότι τοπικές λύσεις μπορεί να υπάρχουν και όλοι πρέπει να ξαναδούμε την επιστροφή στη φύση και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Οι νέες χώρες που κάνουν τα ίδια λάθη που κάναμε εμείς, ίσως μπορούν να προβλέψουν την καταστροφή. Γιατί παραδείγματο χάρη υπάρχουν και άλλα ποτάμια και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Θεωρώ ότι το δικό σας πρόγραμμα είναι μια πολύ καλή ιδέα και ότι σαν Ευρωπαίοι πρέπει να δεσμευόμαστε όλοι. Όταν ε, έρχεται κανείς σε επαφή με τους νέους, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για την εθελοντική εργασία των νέων. Και σε αυτή την περίπτωση και σε 46 χώρες της Ευρώπης δίνεται δυνατότητα εθελοντικής εργασίας στους νέους. Αυτό λοιπόν που εσείς κάνατε σε ένα περιορισμένο πλαίσιο, ίσως υπάρχουν δυνατότητες να επεκταθεί και σε ένα ευρύτερο πεδίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω να συνεχίσετε με μεγάλη όρεξη τα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα και σχέδια που έχετε ξεκινήσει. Εμάς τουλάχιστον μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεχίζουν να υπάρχουν τόσο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ πολύ bedeutet, dass wir, dass sie Όσον αφορά την έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών, δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Α, ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εδώ κυρία Μπαϊ από το Σοσιαλιστές, αλλά συμφώνησα μαζί της να προτείνω για την επίσκεψη που αντιστοιχεί στην χώρα που έχει την Προεδρία, στην Ισπανία που αναλαμβάνει την Προεδρία το επόμενο εξάμεινο. Ήταν η Καταλωνία η ιδέα μας η αρχική. Δεν ήταν τόσο η Βαρκελόνη αυτή καθεαυτή, αλλά πολιτιστική κληρονομιά που είναι εκκλησίες που έχουμε στην Καταλωνία. Τη Βαρκελόνη όντως την έχουμε επισκεφθεί ήδη. Οπότε θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε ένα άλλο σημείο στην Ισπανία. Εγώ βρίσκω ότι θα ήταν καλό να ακούγεται η γνώμη των Ισπανών Ευρωβουλευτών εδώ, από την κυρία Μπαΐα, εγώ και ο κ. Ζερμιγιάν που είναι αναπληρωματικός δεν λέμε ότι έχουμε τίποτα εναντίον του Σαν Σεμπαστιάν, που φυσικά είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ισπανίας, αλλά δεν πρόκειται τόσο για πόλη, πρόκειται να αποφασίσουμε τι θα δούμε εκεί που θα πάμε. Γι' αυτό και θα θέλαμε αυτό να το αφήσετε σε μας και να σας κάνουμε εμείς καινούργια πρόταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, το συζητήσαμε επί μακρόν και διαπιστώσαμε ότι έχουμε πάει πολλές φορές στη Βαρκελόνη. Προηγούμενη θητεία, πέρσι και ότι ίσως καλό θα ήταν να πάμε και σε καμιά άλλη περιοχή της Ισπανίας. Η Ισπανία λοιπόν έκανε αυτή την πρόταση την οποία συζητήσαμε, ψηφίσαμε χτες το βράδυ. Μπορούμε αν θέλετε να ξαναψηφίσουμε αλλά νομίζω ότι η πρόταση να πάμε στο Σαν Σεμπαστιάν θα πρέπει να την ε, ε, κρατήσουμε. Ίσως το 2016 να γίνει και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Δεν λέω, η Βαρκελόνη πάντα έχει πολλούς λόγους να μας προσελκύσει, αλλά έχουμε πάει πολλές φορές στη Βαρκελόνη. Γι' αυτό και χτες σκεφτήκαμε να ακούσουμε και την άλλη ισπανική πρόταση και να πάμε στο Σαν Σεμπαστιάν. Σας παρακαλώ, ας μην επιμείνουμε προς το παρόν, μην επιμείνετε τουλάχιστον για τη Βαρκελόνη εσείς, το σκεφτήκαμε χτες, βέβαια αν επιμένετε θα ψηφίσουμε. Δεν επιμένω για τη Βαρκελόνη, εγώ γι' αυτό για το οποίο επιμένω είναι κάτι άλλο. Η πρόταση που συζητήσατε χτες για το Σα Βαστιέν δεν προέρχεται από την Ισπανία, αλλά από τους φιλελεύθερους που δεν έχουν κανέναν Ισπανό. Οπότε δεν είναι πρόταση που έρχεται από τους Ισπανούς. Ο κύριος Τάκουλα την έκανε χτες από την Φιλενδία, φιλελεύθερος. Με κάθε σεβασμό που έχω απέναντι στο άτομό του. Ωραία, να αποκλείσουμε τη Βαρκελόνη, εγώ δεν λέω. Αλλά ακούστε με τι άλλο την κυρία Μπαγία και εμένα που είμαστε Ισπανοί γιατί στο κάτω-κάτω εμείς θα οργανώσουμε αυτό το ταξίδι που θα γίνει στην Ισπανία. Οπότε αφήστε μας να αποφασίσουμε και σας λέω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα εγώ δεν μπορώ να εγκρίνω αυτή την πρόταση για το Σαν Σεμπαστιάν. Για το ίδιο θέμα θέλετε να πάρετε το λόγο. Λοιπόν, εχθές το απόγευμα αποφασίσαμε. Μπορείτε βεβαίως να επανέλθουμε. Κυρία Χάνιμπολ ήσασταν παρούσα χτε. Μπορούμε αν θέλετε να το ξανασυζητήσουμε στην επόμενη ημερήσια και να πούμε θα πάμε στην Ισπανία και θα δούμε πού θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση πού ακριβώς θα πάμε στην Ισπανία. Βεβαίως και αφορά τους Ισπανούς συναδέλφους το θέμα αυτό και εγώ είχα καταλάβει ότι πρόκειται για ισπανική πρόταση, γι' αυτό και την υποστήριξα. Αλλά Κοιτάξτε, επειδή εδώ υπάρχουν μόνο άτομα από την Καταλωνία, ίσως θα πρέπει να ακούσουμε και κάποιους εκπροσώπους άλλων περιοχών. Η κουλτούρα και ο πολιτισμός στην Ισπανία δεν είναι μόνο καταλωνική. Γι' αυτό και δεχτήκαμε το Σαν Σεμπαστιάν. Μάλιστα ακούσαμε και το όνομα στα Βάσκικα, το οποίο και δεν το γνώριζα. Εν πάση περιπτώσει. Όλοι συμφωνούν να πάμε στην Ισπανία. Το πού θα πάμε θα το ξανασυζητήσουμε. Σε ποια πόλη θα πάμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά των συντονιστών. Για τα πρακτικά της χτεσινής συζήτησης. Ή κάτι άλλο θέλετε να πείτε. Για τους συντονιστές. Ναι, έχετε το λόγο. Ε, ε, e, Επιτρέψτε μου Λοιπόν, να πω ότι ένα, μια ακρόαση για τα πνευματικά δικαιώματα ε, θα ήταν σημαντική και η Πρόεδρος το ανέφερε σε σχέση με το Google μήπως πρέπει να το αναβάλουμε για το 2011 όμως γιατί η Επιτροπή μας από την άποψη της ε, εισαγωγή των δικαιωμάτων ε, των πνευματικών θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να, διερωτη... να ρωτήσω γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί. Δεν ξέρω για το 2011. Αυτό που ξέρω είναι ότι η νομική επιτροπή και η δική μας θα οργανώσει μία ακρόαση για το θέμα αυτό. Από κοινού. Το θέμα του copyright αφορά τη νομική το περιεχόμενο αφορά εμάς, αλλά ίσως